Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ ας αρχίσουμε. Συνάδελφοι, θα ήθελα λίγη ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα. Α, γιατί θα σας πω μια πολύ θλιβερή είδηση, μια συντριβή αεροσκάφους αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Γαλλία. Αεροπορική τραγωδία με πολλά θύματα. Δεν ξέρουμε με ακρίβεια τον αριθμό τους. Νομίζω ότι μπορούμε, χωρίς να περάσουμε σε λεπτομέρειες, να κρατήσουμε αμύτη άλλο ενός λεπτού σιγή για την αεροπορική τραγωδία στη Γαλλία σε συμπαράσταση προς τους Γάλλους συναδέλφους. Παρακαλώ, ενός λεπτού σιγή. Thank you very much. Uh, <clears throat> Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 15. Μελλοντικά μέτρα πολιτική στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος. Ανταλλαγή απόψεων με τον Μιγέλα Ριασκανιέτε, Επίτροπο για τη δράση στο κλίμα και την ενέργεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε τον Επίτροπο Νιγελαρία Κανιέτε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε την ιδιότητα του Επιτρόπου, γιατί ε, πριν από 20 χρόνια ήταν Ευρωβουλευτή. Εγώ βέβαια δεν ήμουν τότε Ευρωβουλευτή, αλλά φαντάζομαι κάποιοι από του παρόντε σα θυμούνται από τότε. Ο Επίτροπος ε, Αρίας Κανιέτε σε άτυπη συνάντηση που είχαμε με την Ήτρη στις 10 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο ε, μας παρουσίασε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση της ε, διασύνδεσης, της διαλειτουργικότητας, πολύ σημαντικό θέμα και είμαστε έτοιμοι να συντάξουμε και έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, για το θέμα αυτό. Δεν αποφασίσαμε ακόμη τις λεπτομέρειες, αλλά θα γίνει μάλλον. Τότε ε, συζητήσαμε αυτό το θέμα και τώρα θα συζητήσουμε τις μελλοντικές ε, πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Μετά την πρόσφατα υιοθετηθήσα στο Συμβούλιο ε, Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Θέμα ζωτικής σημασίας για όλους μας. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας ε, την θλίψη και την προσωπική μου αλλά και τη λύπη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που έγινε το πρωί στις Γαλλικές Άλπεις και θα ήθελα να στείλω τα θερμά μου συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, δέσμευσή του, το σχολιασμό του και την υποστήριξη της Ενεργειακής Ένωσης. Βέβαια, τα λόγια δεν αρκούν για άνθρωπους ε, που θα έχουν να ε, πληρώσουν την θέρμανση και τους λογαριασμούς τους για την ενέργεια. Το στρατηγικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση θέτει το βασικό πλαίσιο για το μέλλον και με τη στρατηγική αυτή θέλουμε να δώσουμε συνοχή στις πράξεις μας και να περάσουμε σε μια νέα φάση ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτό το φω σήμερα θα επικεντρωθώ στην ανταλλαγή απόψεων στις συγκεκριμένε δράσεις αυτής της στρατηγική. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να μιλήσω για τα πρώτα βήματα αυτού του σχεδίου δράσης, ε, τι διασυνδέσεις. Όπω ήδη γνωρίζετε, η ανακοίνωση με το στόχο του 10% του ηλεκτρισμού στο στόχο της διασύνδεσης υιοθετήθηκε ταυτόχρονα με το έγγραφο για την Ενεργειακή Ένωση. Ε, βέβαια, 12 χώρες μέλη ακόμη κάτω το 10% του στόχου αυτού για τον ε, ηλεκτρισμό. Και ελπίζουμε μέχρι το 2020 να διορθώσουμε την κατάσταση στην αγορά ηλεκτρισμού. Χαίρομαι για τις ε, πρόοδους των τελευταίων ετών ε, χάρη σε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στις ενεργειακές υποδομές. Μάλιστα, με τον κανονισμό TNT θα υιοθετήσουμε προγράμματα κοινού συμφέροντος και μαζί με το Συνδέοντας της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαψή για την Ενέργεια θα ε, σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Με το νέο πλαίσιο έχουμε ήδη αποτελέσματα. Η ε, το SLIM 2, η διασύνδεση με την Εστονία και ο άξονας διασύνδεσης Γαλλίας-Ισπανίας είναι σαφή παραδείγματα αυτής της πρόοδου. Την περασμένη εβδομάδα στην Μαδρίτη μίλησα για, την ε, για το διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου και ο κύριος Αυτσόβης μας ε, ενημερώσε για, την, για το φυσικό ε, αγωγό που περνάει από την Ανατολία. Έτσι θα διαφοροποιήσουμε την προμήθεια φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασμού. 10 ε, εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο θα έχουμε πλέον. Χρειάζεται όμως περισσότερη δράση, δηλαδή καλύτερη συνεργασία και συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες επενδύσεις και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Και μέχρι το 2020 εδώ όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν υιοθετήσει το στόχο του 10% διασύνδεσης, με δύο εξαιρέσεις. Ε, η Κύπρος εξακολουθεί ε, να είναι νησίδα αν ε, μέχρι το 2023 δεν ολοκληρωθεί ο σχετικός αγωγός και η Ιβηρική Χερσόνησος επίσης θα ξεφύγουν από την απομόνωση Ελπίζοντα ότι θα περιλάβουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο κοινό μα σύστημα και δημιουργώντα άξονε μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μάλιστα θα έχουμε και ένα νέο, ε, μια περιφερειακή ομάδα υψηλού επίπεδου και αυτό το ανήγγειλε πριν από λίγε εβδομάδε ε, στη διάσκεψη τη Μαδρίτη, ο πρόεδρο Ιούνκερ. Μάλιστα, μέχρι τα μέσα του έτου θα έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα. Επίση, ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία στην Νότια Ευρώπη και στη Βαλκανική Χερσόνησο. Και μάλιστα θα πρέπει να ενισχύσουμε όλες τις περιφερειακές ομάδες ε, και να υιοθετήσουν τις προτεραιότητες για τα ενεργειακά θέματα. Θα σας ενημερώνω πιο λεπτομεριακά και τους επόμενους μήνες για όλα αυτά τα σχέδια. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, πρέπει η εντολή μου τον Οκτώβριο του 2013 και τον Μάρτιο του 2015 για την ε, στην δήλωση για την Ενεργειακή Ένωση θα έχουμε μια δυναμική διαδικασία εφαρμογής της Ενεργειακής Ένωσης. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία διακυβέρνησης και παρακολούθησης ώστε σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό να συνεργαζόμαστε για τον ίδιο στόχο. Θέλουμε ε, ελαστική και υπεύθυνη αλλά και υπόλογη διακυβέρνηση με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης για, το, για την Ενεργειακή Ένωση. Καταρχήν το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται από την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Και μάλιστα μετά τα τεστ αντοχής για την ενεργειακή ασφάλεια και την ε, στρατηγική ασφάλειας ε, θα υποβάλω μέχρι το τέλη του 2015 ένα πακέτο που θα απαρτίζεται από πολλά στοιχεία. Κυρίως μια πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια ε, προμήθειας ε, φυσικού αερίου σε περίπτωση διαταραχής της προμήθειας και θα ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρακολούθηση και τη διαχείριση της κρίσης προμήθειας. Επίσης θέλουμε να αξιοποιήσουμε ε, το δυναμικό μας για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, υποδομές μεταφορών. Θα πρέπει να άρουμε τις, τους φραγμούς για την εισαγωγή τέτοιου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες και άλλους προμηθευτές. Η ενεργειακή ασφάλεια αφορά και τον ηλεκτρισμό. Και υπό αυτό, αυτή τη σκοπιά θα υποβάλουμε νομοθετικά μέτρα για την ε, ενεργειακή ασφάλεια στον ηλεκτρισμό το 2016. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενιαίες προδιαγραφές για την ενεργειακή ασφάλεια του ηλεκτρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πρώτα μια αξιολόγηση της ασφάλειας στην προμήθεια ηλεκτρισμού. Και τέλος, ασφάλεια σημαίνει και ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, την θέσπιση ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με τι κυβερνητικέ συμφωνίε μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Και θα υποβάλω μια πρόταση αναθεώρηση τη σχετική απόφαση για το 2016. Μια ανταγωνιστική και ασφαλή ενεργειακή αγορά θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά τη Ενεργειακή Ένωση. Θέλουμε και hardware πιο ισχυρό και πιο διασυνδεδεμένο, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και μια γνήσια, αυθεντική εσωτερική αγορά στην οποία θα εφαρμόζεται πλήρως η ενωσιακή νομοθεσία. Οπότε θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά το τρίτο ενεργειακό πακέτο, κυρίως σε σχέση με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Από τη στιγμή που εφαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε και ως άμεσα μέτρα θα υποβάλω μια πρόταση για την ενίσχυση της λειτουργίας των NCOs για το 2015 και 2016. Και ο ρόλος της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ε, ήταν θεμελιώδης για την ε, ενσωμάτωση του ενεργειακού και εκτιμένου της Ένωσης και θα συνεχίσουμε τον εντατικό μας διάλογο. Ευχαριστούμε βουλευτές. Η ενεργειακή χρήση αποτελεσματικής συνεργασίας είναι το επόμενο θέμα στην θεματική μας, οπότε για να ξεκαθαρίσουμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή φέτος πρόκειται να προκύψει η στατική μα, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιε δυνατότητες μα. Επίσης θέλουμε το, η κατοθεσία και σχετική νομοθεσία να αναθεωρηθεί, ούτω ώστε να ταιριάζει σκοπούς μα, το 2016 πρόκειται να παρουσιάσουμε μια αναθεώρηση της οδηγίας για την αποτελεσματική χρήση της και πρόκειται κατόπιν να έχουμε μια οδηγία όσον αφορά τα, την αποτελεσματική χρήση στα κτίρια. Το ΣΤΕΚΤ επίση θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, το μετασχηματισμό σε συγκεκριμένα μέτρα τον Οκτώβριο. Και οπότε με την αναθεώρηση αυτή τη οδηγία θα έχουμε και κάποια πρόταση για να τροποποιηθεί το άρθρο Τρία, όσον αφορά τους στόχους της αποτελεσματικότητας για να προσαρμοστεί στο στόχο του 2020 και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μας είπε ότι θα πρέπει με το 2020 να γίνει αυτή η αναθεώρηση έχοντας υπόψη ε, αυτό το, το, το στόχο του 3% για όλη την Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε, τόσο να είναι πιο αποτελεσματική η ενέργεια στην Ευρώπη, να είναι πιο αξιόπιστο, πιο βιώσιμο, γιατί αυτό ε, μετράει για την καθημερινή ζωή των πολιτών από πλευρά εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει σημασία για το κόστος που πληρώνουμε για την ενέργεια και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Και οπότε προβληματιζόμαστε για το πώς θα γίνει κάτι λειτουργικό, αυτό το πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα, να, αποφύγουμε να βρούμε κάποια απόφαση. οπότε ε, αυτή η πολιτική για το κλίμα είναι φιλόδοξη για να έχουμε οικονομία χωρίς ε, άνθρακα και βασίζεται στους στόχους του 2030 οπότε θα πρέπει και έτσι αποφασιστικά να μπούμε στο μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομίας χωρίς άνθρακα αλλά έτσι να έχουμε ανταγωνιστικότητα βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση οπότε ε, αυτό το οποίο κάνουμε ε, εντάσσονται στο πρόγραμμά μας για το 2015. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για την σταθερότητα της αγοράς, να έχουμε αναθεώρηση της οδηγίας για τις ποσοστώσεις των εκπομπών και κατόπιν να δούμε πώ θα γίνει η μείωση των εκπομπών ε, σε σχέση με το σύστημα που υπάρχει το ETS. Και είπαμε ότι μέχρι το 2030 να έχουμε μείωση κατά 43% σε σχέση με το 2005 Οπότε υπάρχουν κάποιε κατευθυντήρε για το πού θα εστιάσουμε την προσοχή μα για την υλοποίηση τη πολιτική για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Οπότε να συνεχίσουμε την ε, δωρεάν διάθεση ποστώσεων στην βιομηχανία και κάποια επιδόματα ούτω ώστε να εξυγχρονιστεί η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Τόσο αφορά τώρα τι δηλώσει που αναφέραμε το 2020 έχουμε κάποιους κανόνες για προστασία της βιομηχανίας, ναι. για αυτή τη διάθεση ποσοστώσεων και όσον αφορά το δικαίωμά τους να είναι επιλέξιμοι για, για επιδοτήσεις και θα πρέπει όμως να υπάρχει προστασία και στο μέλλον σε εκείνους τους κλάδους βιομηχανίας που πρέπει κατόπιν της απόφασης του Οκτωβρίου του 2014. Παρ' όλα αυτά όμως να μην ξεχνούμε ότι τα, τα περιθώρια αυτά και είναι περιορισμένα και άρα θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των επιτρεπμένων προστώσεων. Οπότε έτσι θα πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική και καινοτόμα βιομηχανία. Και αποφασίσαμε να συνεχιστεί το τρέχον σύστημα. Οπότε και το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ισχύει το benchmarking. Αυτή η το σύστημα προστασία για τις διαρροές καθώς, και η διάθεση των προστώσεων. Επίσης εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι απόψει των εμπλεκομένων οπότε είναι ε, καλοδεχούμενε οι τύχουν προτάσεις σε σχέση με το ETS. Πέραν του ETS εμείς ξεκινήσαμε μια προπαρασκευή για κάποιε νομοθετικέ πρωτοβουλίε για του τομεί e εκτό του ETS, εκτό Ευρώπη, Οπότε να έχουμε επίπτωση μελέτη επιπτώσεων και επίσης διαβουλεύσεις. Θα προκύψουν αποφάσεις κατά το πρώτο του 2016. Επίσης, οι στόχοι εκπομπών σε εθνικό επίπεδο θα ακολουθήσουν και θα συνδέονται και με το, το κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με το ΑΕΠ, ώστε να έχουμε ε, μια ρύθμιση με καλή σχέση κόστους αποτελέσματος. Οπότε θα πρέπει να αποκτήσουμε και μια αγορά για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ε, ενέργειας. Οπότε θα πρέπει η σχετική οδηγία να αναθεωρηθεί για την περίοδο μετά το 2020 και έτσι να αντιμετωπίσουμε μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που έχουν σχέση με την ολοκλήρωση της αγοράς για την ανανεώσιμη ενέργεια. Οπότε θα κατεβάσω σύντομα μια δέσμη μέτρων. Νομοθεσία για να πετύχουμε τους στόχους 2030, και να έχουμε έτσι ε, με χαμηλό κόστος μια νέα πολιτική. Ε, και έτσι να είμαστε πρωτοπόροι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μπορούμε ε, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οπότε έχουμε το σχετικό πρόγραμμα δράσης που θα δημοσιοποιηθεί με το τέλος του 2015 οπότε και θα αναλύσουμε στο πώς έχει τώρα το τοπίο, το τεχνολογικό και τι πρέπει να κάνουμε. Θα κλείσω κυρίε και κύριε κάτι το οποίο υποψιάζομαι ότι θα μου θέσετε. Σχετικά με την μεταβολή του κλίματος. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, λήψη και αποθεματοποίηση του άνθρακα. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο να έχει σχέση με το σύστημα εμπορίας των ποσοστώσεων. Περιμένω πάντως τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την ε, εισηγήσή σας. Πάρα πολύ σφαιρική και καλύψατε πάρα πολλά ζητήματα νομοθετικά και μη νομοθετικά όμως όσον αφορά την πολιτική την ενέργεια και το κλίμα. Πρώτα πρώτα λάβουν το λόγο οι συντονιστές μας και πρώτος είναι ο κύριος Κάρινς. Τρία λεπτά. Συγγνώμη που σα διακόπτω κύριε Κασιάνης. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, εντάξει, τότε θα μιλήσω πιο πολύ για να καλύψω το διάστημα των τριών λεπτών. Ο κύριο Κάριν. Μία ερώτηση κατευθείαν να θέσω. Σω δεν τα καταφέρω. Μιλήσατε για του αγωγού διασύνδεση. Ε, ότι 12 καρδιμέλοι είναι κάτω από το στόχο αυτό. Σε ό,τι αφορά τα κατασκευαστικά έργα για τη βελτίωση της κατάστασης. Η ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι η εξή. Όταν θα υπάρχουν ε, φυσικά η φυσική αγωγή, πόσο θα απέχουμε ακόμα από μια λειτουργούσα αγορά. Ποια είναι τα εμπόδια που υφίστανται σήμερα σε ό,τι αφορά τα εθνικά δηλαδή εμπόδια που υφίστανται. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία για το για την διασύνδεση, όχι μόνο η αγωγή. Ως νομοθέτης λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε για να άρουμε τα εμπόδια αυτά, προκειμένου αυτό το 10% διασύνδεσης να έχει νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Dan Ευχαριστώ και επίτροπε, σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το σχέδιο δράσης αυτό καλωσορίζουμε το σχέδιο δράσης. Και θα θέλαμε καταρχάς να καλωσορίσουμε τη συνοχή των όσων μα είπατε και επίσης τη συνοχή με αυτά που μα είπε και ο κ. Σεύκοβιτ σε ό,τι αφορά θέματα διασύνδεση. Αυτό που καμιά φορά μας προκαλεί ανησυχία είναι το εξή. Ο στόχος αυτός για το 2020 θα πρέπει να υπάρχει ετήσια έκθεση προκειμένου να καταγράφεται η πρόοδος ανέτος, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές αν μέλος σε ό,τι συμβαίνει. Κατά δεύτερον, όταν μιλάμε για ανταλλαγέ ηλεκτρικού αερίου κτλ. από τις διάφορες χώρες, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση αυτών των ροών Ύστερα θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει. Ε, για παράδειγμα υπάρχει ήλιος ε, στον νότο της Ευρώπης. Θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε την ενέργεια αυτή. Και αντίστροφα σε ό,τι αφορά την, ενέργεια θέρμανσης. Όλα αυτά δεν έχουν διελευκανθεί. Πώς θα μεταφερθεί δηλαδή η ενέργεια από τον βορρά στο νότο και τον νότο στο βορρά. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Μιλάμε για τη διαφοροποίηση των παραγωγών για την ε, μετακίνηση από την Ανατολή στη Δύση. Ίσως αυτό να αποτελεί μια ένδειξη ότι τα πράγματα στο μέλλον θα τα πάρουμε πιο σοβαρά. Είναι καλό αυτό το σημάδι. Και κάτι που θα ήθελα να καλωσορίσω, αυτό που είπατε για τις ανανεώσιμες. Αυτό φαίνεται ότι το λαμβάνουμε πολύ πιο πολύ υπόψη πλέον. Η βιομηχανία αυτή, ο κλάδος αυτός χρειάζεται υποστήριξη και όχι μόνο στα χαρτιά, πραγματική υποστήριξη προκειμένου να αναπτυχθεί. Θα γίνουν λοιπόν πιο πολλές επενδύσεις στην έρευνα για τις ανανεώσιμες και αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος αυτός θα αναβαθμιστεί. Γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι είναι λίγο δύσκολη πηγή ενέργεια, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ότι δεν είναι αξιόπιστε και το καθεξής Και νομίζω ότι το πακέτο για τι ανανεώσιμε θα δώσει μια όθηση στον κλάδο αυτό. προκειμένου να μειωθεί, αν θέλετε, ο απρόβλεπτος παράγοντας. Και τέλος, ένα τελευταίο στοιχείο σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για τη διάσκεψη του Παρισιού. Πώς θα ενημερώσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το ότι συμβαίνει στο Παρίσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ΕΛΚ, ήταν ο πρώτος ομιλητής από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, ο δεύτερος από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές λίγο αργότερα και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Φέντερλε από την Άλτε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ και χαιρόμαστε που βρίσκεται βρίσκεται μαζί μας. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή τη θητεία. Μια μεγάλη ευκαιρία για μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική η οποία θα έχει πιο επικοδομητικό χαρακτήρα από ό,τι στο παρελθόν. Μιλάμε για το πετρέλαιο, για τον άνθρακα, για το αέριο, αλλά το είπε αυτό και προηγούμενος συνάδελφος. Περιλαμβάνεται και ανανέωση μέσα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Μεγάλα ποσά δίνονται ανά ημέρα ακόμα. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόθεση των ορευτών καυσίμων που είναι αρκετά επιζήμια για το περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καλή αίσθηση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με εσά εδώ κύριε Επίτροπε Καλνιέτε. Δεν είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τα ορυκτά καύσιμα, τη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει μια παράλληλη στρατηγική, παράλληλη ανάπτυξη, παράλληλη ε, ανάπτυξη τέτοιων τρόπων παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό ότι και ο άνθρακας παρέχει δυνατότητε ανάπτυξης και οικονομική ανάπτυξης, αλλά να λάβουμε υπόψη και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Να επικεντρωθούμε πιο πολύ λοιπόν στις ανανεώσιμες για το μέλλον. τα πράγματα διαφέρουν ανάλογα με την ενεργειακή κουλτούρα τη κάθε χώρα στην Ευρώπη. Θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση με τον τρόπο αυτό. Πολλά δεν λειτουργούν άρεστα στην έννοια αγορά. Και αυτό φυσικά θα έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον ενεργειακή πόρη που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν Οπουδήποτε στην ε, Ευρώπη για τα πλεονάσματα υπάρχουν κανόνες και πρόκειται για μεγάλη σπατάλη πόρων γιατί έχουμε ενεργειακό πλεόνασμα σε πολλά μέρη στην Ευρώπη. Εγώ είμαι Σουηδός. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε προκειμένου να βρεθεί μια ενεργειακή λύση στη Βαλτική σε ό,τι αφορά αγωγούς μεταξύ Βαλτικής και Βορρά. Υπάρχουν τέτοια σχέδια τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν για την ενεργειακή πολιτική και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια κοινή βάση για τις εργασίες αυτές με τους συναδέλφους από την Επιτροπή. Ψηφίσαμε άλλωστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας και για το και το αεροπορικών ε, αεροπλοίας και σε όλες τις συζητήσεις αυτές ουσιαστικά επαναρχόμαστε στο ίδιο σημείο, πράσινες αναλλακτικέ. Ενώ σημαίνουν τα αντίθετα ουσιαστικά, χρειαζόμαστε μια πολιτική λοιπόν ανταπόκριση Ρωτώ λοιπόν στον Επίτροπο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μελλοντικά αυτή τη στρατηγική προκειμένου να υπάρχουν και οι δύο πλευρές και να μην υπάρχει αντίφαση. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανομή της ενέργειας. Ευχαριστώ ο Κλόπ Τουρμής από τους Πράσινους που ποτέ δεν κάνει, δεν χάνει χρόνο. Πάντα δραστηριό. Έχετε το λόγο, Κλοντ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μόλι με ενημέρωσαν για την ομιλία σας. Χαίρομαι που μας παρουσιάσατε όλες αυτές τις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σας. Κάτι που επισήμανα και, στον, και που θα επισημάνω αύριο στον Επίτροπο, μάλλον χθε επισήμανα στον Επίτροπο Σεύτσοβιτς, είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά. Υπάρχει όμως σήμερα τεράστια στρέβλωση στην ενιαία αγορά εξαιτία των επιχορηγήσεων και μη εσωτερήκευση των εξωτερικών παραγόντων. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια εκτεταμένη έρευνα και κατέληξε στη μελέτη κοφή το Δεκέμβριο. Μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες λεπτομέρειες της μελέτης, αλλά τα βασικά συμπεράσματά της είναι το εξής. Στην εσωτερική αγορά η μεγαλύτερη στρέβλωση γίνεται υπέρ των ορυκτών καυσίμων. Στη συνέχεια υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και μόνο ε, στην τρίτη θέση έρχονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που βλέπουμε τώρα και ακούμε είναι το επιχείρημα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά στην αγορά. Κανένας δεν είναι αντίθετος. Αλλά αν η αγορά δεν φτιάχνονται γύρω από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, οι τιμέ του δεν θα είναι προσιτέ. Η ενεργειακή αγορά σήμερα δεν είναι φτιαγμένη, δεν είναι σχεδιασμένη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αγορά ενέργεια ε, σχεδιάστηκε στις αρχές τη δεκαετία του 90 για εργοστάσια που ουσιαστικά αγοράζουν ενέργεια, δεν παράγουν ενέργεια. Οπότε δεν είναι προσαρμοσμένη η αγορά μας στις ανάγκες των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις τρευλώσεις στην αγορά ενέργειας. Και κάτι που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό είναι ότι στη Γερμανία που έχουμε ίσως τις πιο σταθερές καταστάσει και την πιο διεξοδική νομοθεσία, οι επίσημες ε, πηγές από το Υπουργείο λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια της Γερμανίας. Ε, το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί ότι θα ενέκυπτε αυτό το θέμα. Και ακριβώς επειδή δεν ασχολήθηκε, το 2004 η British Energy χρησιμοποίησε, σε άλλους σκοπούς τα τεράστια κονδύλια που έχει συγκεντρώσει για τον παραπλησμό των πυρηνικών εργοστασίων. Τι θα γίνει, θα μετακυλήσουμε στους φορολογούμενους όλο το κόστος που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει οι διαχειριστές των πυρηνικών εργοστασίων και εδώ δεν είναι αν κανείς υπέρ κατά της πυρηνικής ενέργειας. Θέλουμε μια δικαιοσύνη στην αγορά ενέργειας. Και οι παραγωγοί θα πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος, όχι οι φορολογούμενοι. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Τώρα, ο κύριος Νεοπλής Ηλικιώτης. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, το πρώτο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι σε σχετικά με την απομόνωση κρατών μελών και περιοχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Είναι γνωστό ότι και προς και Μάλτα, πολλά νησιά, πολλές ορεινές περιοχές είναι απομονωμένα ε, περιοχές. Ο στόχος για να αρχίσει αυτή η απομόνωση που τέθηκε για το 2015 δεν φαίνεται να υλοποιείται. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί εκ των πραγμάτων. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει στους σχεδιασμούς η προοπτική ε, για την άρξη της απομόνωσης αυτών των κρατών πέραν από κάποιες γενικές αναφορές. Το δεύτερο, μιλήσατε για ολοκληρωμένη στρατηγική υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ε, ενώ υπάρχουν στα σκαριά ε, πολιτικές για στήριξη, για δημιουργία σταθμών ε, από υγροποίησης ε, και στην περιοχή της Μεσογείου Εκείνο που απουσιάζει είναι να δούμε μια α, θέση, μια σκέψη, μια πρόταση για στήριξη ε, σταθμού υγροποίηση. Γιατί υπάρχει δυνατότητα ε, στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου να δημιουργηθεί σταθμό υγροποίηση ο οποίο να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Το τρίτο θέμα, όπω γνωρίζετε, ε, οι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου ε, έχουν αντιμέτωπε με έναν ιδιαίτερα ψηλό κίνδυνο σε περίπτωση που δημιουργηθούν πυρηνικοί σταθμοί στην περιοχή. Και αναφέρουμε, σχεδιάζεται να αναγερθεί πυρηνικό σταθμό στο Άκιο τη Τουρκία, καθώ και μεταφορά πυρηνικών αποβλήτων που εγκυμενούν σοβαρού κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αποτελεί δε σοβαρή απειλή και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονό ότι πρέπει να λάβουμε την υπόψη ε, τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ατυχήματο, λαμβάνοντα υπόψη ότι μιλούμε για μια σεισμογενή περιοχή, ίσω από τι πιο σεισμογενείς περιοχέ ε, στο, στον κόσμο. Το ερώτημα κύριε Επίτροπε είναι ποιε ενέργειε θα προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή ε, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην περιοχή της Ανατολική Μεσογείου ε, και να υπερασπιστεί ιδιαίτερα τα δικαιώματα στην ασφάλεια κρατών μελών όπω είναι η Κύπρο, η Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποτραπούν τα σχέδια τη Τουρκία η οποία ω γνωστόν είναι μια υποψήφια για ένταξη χώρα ε, να αποτραπεί από το να δημιουργήσει πυρηνικό σταθμό σε μια επικίνδυνη και σεισμογενή περιοχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ. Ίσως αργότερα έρθει εκπρόσωπος ε, της EFDD. Ολοκληρώσαμε το γύρο των συντονιστών και θα ζητήσω από τον κύριο Επίτροπο να απαντήσει τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ξεκινήσω με τη δύσκολη ερώτηση που υπέβαλε εκπρόσωπος ε, του ΕΛΚ για τις διασυνδέσεις. Είναι πολύ καλός ο στόχος, αλλά μετά τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο, στο σχεδιασμό της αγοράς. Γιατί οι γραμμές διασύνδεσης είναι το hardware, θέλουμε και software, θέλουμε φιδίκτυα παντού. Επίσης, να καταργήσουμε τις τρευλώσεις ε, της ενέργειας και να ενισχυθεί η ικανότητα πληρωμών. Γιατί αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο και έχουν διαφορετικά συστήματα ε, ικανότητων. Και αυτό θα στο μάλλον θα δημιουργήσει δυσκολίε. Επίσης, ρυθμιζεμένε τιμέ. Και αυτό είναι ένα, ένα θέμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Γιατί υπάρχουν εμπόδια με τις διαφορέ των τιμών. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον ίδιο το σχεδιασμό τη αγορά. Και αυτό είναι θέμα των ε, εξουσιών του ΕΣΕΡ, του, της Επιτροπής ε, Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών. Να δούμε πώς θα έχουμε την, ε, να διευρύνουμε την εθνική προσέγγιση στις ικανότητες, να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με κοινά καθεστώτα, να δούμε πώς θα στηρίζονται στην αγορά και θα καταργήσουμε τις τρευλώσεις, ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, ελαστικοποίηση της αγοράς που θα πρέπει να προσανατολίζεται στη ζήτηση, να βελτιώσουμε το συντονισμό σε επίπεδο διανομής, να δώσουμε πιο ενεργό ρόλο στους καταναλωτές ε, ε, για τον ηλεκτρισμό και επίσης ε, πώς θα ενισχύσουμε το διασυνοριακό ανταγωνισμό των λιανεμπόρων. Γιατί οι γραμμές διασύνδεσης είναι η ραχοκουκαλιά του συστήματος, αλλά δεν αρκούν. Εύστοχη ερώτηση, λοιπόν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα επιμέρους θέματα. Επίσης, τι συνέχεια θα δοθεί για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την υλοποίηση των στόχων σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα συντάξουμε έκθεση για τις πραγματικές εξελίξεις ε, και την κατάσταση των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πού έγκυται τα προβλήματα, πού υπάρχουν στενοποί και να υποβάλουμε μια νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα θα υποβάλουμε να έχουμε ένα μάλλον ε, φιλόδοξο πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια νέα οδηγία ε, θα έχουμε κατευθυντήρες γραμμές για την ε, κατανάλωση, αναθεώρηση της οδηγίας για τις ΑΠΕ, ανταλλαγή των πρακτικών, συστήματα ενίσχυσης της ενέργειας και δεν αρκεί μόνο η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Δεν αρκεί να προσανατολίσουμε τις ΑΠΕ σε ένα, σε ένα διαφορετικό σύστημα αγοράς. Θέλουμε να στηρίξουμε καλύτερα τις ΑΠΕ στην Ενεργειακή Ένωση γιατί μπορούν να δημιουργηθούν διαφορές του ανταγωνισμού ε, μεταξύ των κρατών μελών. Αν έχουμε μαζικές <coughs> κρατικές ενισχύσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη για τι ανα... ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ίσω δημιουργηθεί στρέβλωση ανταγωνισμού. Θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Θέλουμε ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Και γιατί θέλουμε γραμμέ διασύνδεση, interconnectors. Γιατί δεν μπορούμε να αυξήσουμε την ικανότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια χωρί ε, γραμμέ διασύνδεση. Πώς θα φτάσουμε το στόχο του 27% παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχουμε αρκετούς, αρκετές γραμμές διασύνδεσης. Γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε άλλες χώρες έχουμε περισσότερο ήλιο, αλλά έχουμε περισσότερη αιωλική ενέργεια. Μερικές περιπτώσεις θέλουμε να συνδέσουμε το βορρά με τον νότο, ενώ ακόμη και στο εσωτερικό μιας χώρας είναι δύσκολη μερικές φορές η διασύνδεση βορρά και νότου. Εμείς θέλουμε πλήρη διασύνδεση σε περιφερειακό επίπεδο, στηρίζοντας, σε μία, ε, στηρίζοντας πηγές ενέργειας που θα βασίζονται στην αγορά. Τώρα έχουμε πια πολύ όριμες τεχνολογίες. Ε, σε ορισμένου τομεί άλλου, θα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία για να οριμάσουν οι τεχνολογίες. Πάντως, όλα αυτά θα πρέπει να τα στηρίξουμε και με δημόσια κονδύλια. Μία καλή ερώτηση υπευλήθη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τη στρατηγική μας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Αυτή τη στιγμή έχουμε χαμηλές τιμές ορυκτό καυσίμων και χαμηλές πετρελαϊκές τιμές. Και επειδή πολλέ συμβάσει για το πετρέλαιο συνδέονται με το φυσικό αέριο, έχουν πέσει και τιμέ φυσικού αερίου. Με του νέου κόμβου θέλουμε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμό στον τομέα του LNG. Με τη ΣΥΠΑ συζητούμε το TTIP και το TTIP έχει σημαντικό ενεργειακό κεφάλαιο. Εκεί η ελεύθερη εξαγωγή φυσικού αερίου από τι ΗΠΑ και η αποφυγή των διπλών τιμών θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής υγροποιημένου φυσικού αερίου που είναι ζωτική σημασία για το μέλλον για την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Θέλουμε διαφοροποίηση των δρόμων και των προμηθευτών μας και πολύ σημαντική επιλογή θα είναι του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Γι' αυτό και θέλουμε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα εκπονήσουμε μια ευφυή στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο για να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια του, ενεργεια... του ενεργειακού ανεφοδιασμού και να έχουμε φυσικό αέριο και από τους παραδοσιακούς ε, αγωγούς φυσικού αερίου και μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πάντως είναι σημαντικό να υλοποιήσουμε τέτοια πολιτική. Ο κύριος Τούρμες ε, μας μίλησε για τις επιδοτήσεις που δίνονται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα. Όντως, και μάλιστα αυτή τη στιγμή το σενάριο και οι συνθήκε είναι πολύ ευνοϊκέ, γιατί έχουμε χαμηλέ πετρελαϊκές τιμές και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επικεντρωθούμε στο θέμα του τι γίνεται με τις επιδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα. Και να ξανασκεφτούμε όλη την κατάσταση. Γιατί με βάση τα στοιχεία που έχουμε είναι πάνω από 100 δις. 400 δις ε, είναι οι εισαγωγές και 100 δις ε, οι επιδοτήσεις. Είναι ευνοϊκές συνθήκες λοιπόν να εξετάσουμε τα θέματα τώρα και να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε τους ενεργειακούς μας στόχους. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είναι ευνοϊκό και πρόσφορο το έδαφος για να ξεκινήσουμε την αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό, παρόλο που δεν είναι εύκολο. Τώρα, το θέμα του παροπλισμού του κλεισίματος πυρηνικών εργοστασίων και το θέμα της πυρηνικής ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μία ανακοίνωση για, μια, για ένα νέο προγράμμα, πυρηνικό πρόγραμμα με βάση το άρθρο 40 της Συνθήκης Ευρατόμ. Και μάλιστα αυτό το νέο πρόγραμμα θα δίνει πληροφορίες για την κατάσταση των επενδύσεων στην πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μελλοντικές τάσεις δεδομένου των δικτύπων των τελευταίων πολιτικών και θα υποβληθούν και πρωτοβουλίες όπως κανονισμός ε, ε, του Συμβουλίου για τα επενδυτικά προγράμματα στην πυρηνική ενέργεια και κατευθυντήρες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου του αρμόδιου άρθρου της Ευρατόμ που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, το δικαίωμα διαπραγμάτευση συμφωνιών με τρίτε χώρε για πυρηνικά θέματα. Έχουμε μια νέα κατάσταση που δεν ξέρουμε αν θα είναι προσωρινή ή μόνιμη. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί με τις πετρελαϊκές τιμές έχουμε, ανακύπτουν πολλά ερωτήματα. Ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου και τι θα γίνει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το θέμα των επιδοτήσεων δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί επιδοτήσει δίνονται παντού στον κόσμο. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Επίσης, στέθηκε ερώτημα για τα προβλήματα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της ενεργειακής τους ασφάλειας. Εμείς εξετάζουμε την ενεργειακή ασφάλεια πανευρωπαϊκά σε ορισμένες περιφέρειες τα προβλήματα είναι πιο έντονα, σε άλλες λιγότερα. Τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον νότιο διάδρομο, που τηρεί το χρονοδιάγραμμα TAP και τα NAP. Επίσης θέλουμε γραμμές διασύνδεσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως σύνδεση Βουλγαρίας-Ελλάδας Βουλγαρίας, Ρουμανίας ε, και Σερβίας ώστε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 2020 να επιτύχουν διασύνδεση ηλεκτρισμού 10%. Και στόχος για το φυσικό αέριο είναι να έχουμε τρεις διαφορετικούς προμηθευτές και πλήρη διασύνδεση 10% για τον ηλεκτρισμό αν αναπτύξουμε τις γραμμές διασύνδεσης, τις πολιτικές μας και τη στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, πιστεύω ότι θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν. Και τα τεστ αντοχής είναι χρήσιμα γιατί θα μας δείξουν τα ατού μας και τις αδυναμίες μας. Και με αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, με περισσότερες γραμμές διασύνδεσης και καλύτερη ροή της ενέργειας, θα, ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εκ Το σχέδιο της Ενεργειακής Ένωσης έχει μία δυσκολία. Γιατί πρέπει να παίζει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και για ένα μια ισορροπημένη αγορά θα πρέπει εκ να προωθήσουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Ελπίζω να τα καταφέρουμε στην πενταετία που έχουμε μπροστά μας, όπου θα εργαστούμε εντατικά και άοκνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ ανοιχτή και διαλλακτική και θέλει ειλικρινή διάλογο με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Ένωση. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και για τις παρατηρήσεις σας για τις πολύ σημαντικές δραστηριότητες της Επιτροπής Ήτρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή ε, Ήτρε ένα νέο μέλος, τον κύριο Ερμπάν. Καλώς ορίσατε, οπότε βλέπετε είμαστε ίσως και πιο δραστηρία Επιτροπή. Τον κύριο Εσενίκ αντικαθίσταται αν ε, δεν κάνω λάθος. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Άρης Κανιέτε, σαν συνέπεια της διαχείρισης δικής σας και των συναδέλφων σας στην Ισπανία, το ρεύμα για την Αγγερά είναι 72% περισσότερο από όσο ήταν το 2004, από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη πέραν, αυτών των υψηλών τιμών όμως, οι Ισπανοί έχουμε 30 δις ευρώ χρέος. Το βιόλο είναι και αυξάνει. Σύμφωνα με αυτή την, αυτό το τιμολογιακό έλλειμμα. Και τι γίνεται με τις ανεωρνητικές ενέργειες. Γιατί το πιο ασυγχώρητο και το πιο σοβαρό είναι ότι έχουμε 7 εκατομμύρια Ισπανούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στη λεγόμενη ενεργειακή φτώχεια. Παρ' όλα αυτά τα κέρδη αυτών των μεγάλων εταιριών ε, ηλεκτρισμού στην Ισπανία έχουν ουσιαστικά διπλασιαστεί σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό το μοντέλο και αυτή η ενεργειακή πολιτική μας έφτασε σε αυτό το σημείο και σας ερωτώ γιατί στα σχέδιά σας ποτέ δεν μιλάτε για εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στην ενέργεια. Ποτέ δεν συστήθηκε αυτό. Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την ενεργειακή φτώχεια. Και στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, είναι πολύ ενισχυτικό σήμερα μια έρευνα της Γενικής ότι 8 εταιρείε ηλεκτρισμού συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τον αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη λεγόμενη διαδικασία της Σερβίλης. Αυτό κάνουν τα λόμπι αυτών των εταιριών, Ούτως ώστε οι κανόνες να γίνουν πιο χαλαροί όσον αφορά τους ε, σταθμούς, ε, θερμικούς σταθμούς παραγωγής ε, ηλεκτρισμού. Τι λέτε γι' αυτά, Πρόεδρος. Είπαμε στο δεύτερο γύρο ένα λεπτό ή μισή λεπτό κανονικά. Εσεί πάντω ε, κάνατε την παραθενική σα ομιλία στην Επιτροπή μα, οπότε γι' αυτό και σα άφησα να μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά. Και τώρα κύριε Πιλάρντε Καστίγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καλώ ορίσατε αγαπητέ Επίτροπε για άλλη μια φορά στην Επιτροπή μα. Πού είναι η αρμοδιότητά μα η ενέργεια. Πάρα πολύ εντυπωσιακά είναι αυτό το οποίο μα είπατε όσον αφορά μια ξενάγηση στο τοπίο της ενέργειας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τονίζω γιατί ακριβώς το θέμα τώρα είναι να συζητήσουμε πώς ένας ε, ευρωπαϊο επίπεδο θα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα πέραν των όσων κριτικών έχουν διατυπωθεί. Τέλο πάντων οι κριτικέ είναι και αυτέ θεμητέ. πάντω. Σαν μια πρώτη εισήγηση και μία ε, απάντηση ε, όλα ήταν πάρα πολύ σφαιρικά και πλήρη ούτως ώστε δύσκολο κανείς να βρει ερωτήσεις για νέα, ε, νέα θέματα, νέα ερωτηματικά, νέες σκέψεις. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για τις διασυνδέσεις, τι θα κάνετε, προτίθεστε να συγκρατήσετε κάποια περιφερειακά ευρωπαϊκά ευρωπαϊκά γκρουπ, ευρωπαϊκές ομάδες και ακριβώς πώς σκοπεύετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία όσον αφορά τα ευφύ δίκτυα, δηλαδή να μπορέσετε να ενσωματώσετε την ενεργειακή πολιτική το θέμα των ψήφων την ψηφιακή τεχνολογία. Κέλε. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Κάθε φορά που σας ακούω να μιλάτε, έχω την εντύπωση ότι είστε κάποιο, ο οποίο ξέρετε πραγματικά για τι μιλάει και είσαστε διατεθειμένο να κάνετε και κάτι σε ό,τι αφορά θέματα νομοθεσία. Τρία, τρεις λέξεις κλειδιά. Ασφάλεια, διαφοροποίηση και διασυνδεσιμότητα. Ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ενεργειακή Ένωση. Μια τι θα ήθελα να σας κάνω από αυτόν. Στη δική μου περιφέρεια, Υπάρχει μικρή διασύνδεση για το αέριο και γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της θέρμανσης ε, γίνεται με πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε θεωρώ να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκή βάση. Κατά δεύτερον, αναφερθήκατε στην προτινόμενη νομοθεσία για το ευρωποιημένο αέριο. Σωστή, μου φάνηκε. Και αναφερθήκατε και στα κτίρια. Νομίζω ότι Πρόκειται για ένα βασικό τομέα που πολλά μπορούν να γίνουν. Ένα τομέα κλειδί για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί Αναρωτιέμαι πόσο μακριά θα μπορούσαμε να πάμε για να διασφαλίσουμε τα παστικά σπίτια. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, επίτροπε. Χάρηκα πάρα πολύ που βάλετε στο επίκεντρο την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μπορείτε να αναπτύξετε πιο πολύ τη σύνδεση μεταξύ τη αποδοτικότητα τη ενέργεια και τη ένδυα τη ενέργεια. Ξέρουμε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί μια βασική απάντηση στα ερωτήματά μα και θα πρέπει να θεωρηθεί ω ε, πρώτη πηγή ενέργεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα. 75% των κτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μη αποδοτικά και εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο, μια τεράστια σπατάλη. Και στην ανακοινήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η ενεργειακή ένδυα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ένα συνδυασμό μέτρων, αλλά δεν προτείνεται κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Χτες προτάθηκε αναθεώρηση της πολιτικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα και η κυρία Τάισιν θα συμπεριληφθεί ως Επίτροπος στα θέματα αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδυας. Θα μπορούσατε λοιπόν να αναπτύξετε λίγο πιο πολύ το θέμα της νομοθεσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και το πώς σκοπεύετε να συντονιστείτε με την κυρία Τάισεν για την ενεργειακή ένδυα και ποια θα είναι η συνολική στρατηγική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόφορτ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ Uh, να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για μια ενοποιημένη ενεργειακή αγορά. Αλλά αναρωτιέμαι, αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σχέδια έχει για να ενισχύσει το ΕΙΣΑ για τους πόρους, αλλά και για το κανονιστικό τμήμα, γιατί τα εθνικά TSO σε πολλές περιπτώσεις εμποδίζουν την επιτεύξη των στόχων για το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων στην ε, αγορά της ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, εν συντομία, αναφερθήκατε ότι είναι καλό που το Συμβούλιο έβγαλε συμπεράσματα για μια δυναμική δομή διαχείρισης, διακυβέρνησης. Αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους για το 2030, δεν χρειαζόμαστε μόνο δυναμική δυναμικής ε, διαχείρισης για τους στόχους αυτούς. Εύρωστη πραγματικά διαχείριση. Τι είδου ιδέε έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την δυναμική εύρωστη, στεναρή διακυβέρνηση, διαχείριση, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του 2030. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Ζαντού. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. ακούγοντας συναδέλφους ε, διαπίστωσα ότι έχετε ολόκληρο fan club ε, στην Επιτροπή Ήτρε. Κάτι περίεργο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Όταν μιλάτε για ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους, ε, μας αναφέρετε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι δικαιολογεί θεσμικά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να αποτελούν τη βάση για τις εργασίες όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Γιατί δεν ξεκινάτε στο Συμβούλιο ε, στις δηλώσεις σας, δεν ξεκινάτε από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση, τις ανα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν ε, είναι αυτά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί έχουμε δύο βραχιώνε ε, στην νομοθετική εξουσία. Γιατί το Συμβούλιο έχει μεγαλύτερη νομοποίηση από το Κοινοβούλιο. Επίση, είχαμε τη διάσκεψη κορυφή για του ε, γενεί πόρου, ε, για τον άνθρακα. Υπάρχει όμω τεράστια σύγχυση αυτή τη στιγμή. Μήπω οδηγούμαστε σε μια πανεθνικοποίηση των ενεργειακών πολιτικών και κάθε χώρα διαλέγει στο, στο ενεργειακό τη μείγμα ό,τι πηγή θέλει και πέραν του ηλεκτρισμού ελάχιστα είναι τα κοινά στοιχεία στην ενία αγορά ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, έγιναν κάποιες συγκεχημένες δηλώσεις ε, για το διπλό διακύβευμα σε σχέση με τα άειλα αποτελέσματα της επικείμενης διάσκεψης κορυφής για το κλίμα μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι από το Παρίσι θα πρέπει να βγει ένας οδικός ε, χάρτης ε, συγκεκριμένος και δεσμευτικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, προηγουμένως μιλήσατε για την τιμή του πετρελαίου. Όντως, ε, είναι πρωτοφανείς αυτές οι τιμές πετρελαίου. Βέβαια, είναι και θέμα πολιτικής γιατί Σαουδική Αραβία ε, ήθελε να πατάξει τον ανταγωνισμό από το σχιστολιστικό αέριο και τις ασφαλτόδεις ε, άμμος. Ε, ίσως ε, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να θέσουμε μια ανώτατη τιμή και για το διοξίδιο του άθρακα. Γιατί πολιτικοί είμαστε. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή και από αυτή την άποψη. Ο κύριος Βιντάλ. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζουμε τις αξιόλογες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση μιας ε, πιο αιχμηρής ενεργειακής ε, και κλιματικής αλλαγής. Μέσα σε μια ε, μέρα το Φεβρουάριο είχαμε τρεις ανακοινώσεις για την Ενεργειακή Ένωση, τις Δεσιδέσεις και το πρωτόκολλο του Παρισιού. Επιτέλους έχουμε καινούργιες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα από τα σημαντικά σημεία τη Ενεργειακή Ένωση, για να έχουμε καλύτερο συντονισμό τη ενεργειακή πολιτική είναι η έννοια τη διακυβέρνηση. Βέβαια, μένει κάπω συγκεχημένη αυτή η έννοια τη διακυβέρνηση. Πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να συμφιλειώσουμε στενότερη ενεργειακή συνεργασία με το σεβασμό τη εθνική αρμοδιότητα ε, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματο, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει αυτές τις εθνικές αρμοδιότητες. Σε ό,τι φορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, βλέπω ότι είστε υπέρ μια φιλόδοξη προσέγγιση εν ώψη τη διάσκεψη των Παρισίων. Όλοι συμφωνούμε ότι κλειδί τη επιτυχία του Παρισιού θα είναι όλε οι χώρε και κυρίω αυτέ που εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να αναλάβουν αναλογικούς και δίκαιους στόχους μίας εκπομπών. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα αποτελέσματα των Παρισίων. Έχω όμως μια ερώτηση. Έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αρμόδια για το 9% των παγκόσμιων εκπομπών θα είναι η μόνη που διακόπτει δυστυχώ ε, ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θεωρώ ότι η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί σίγουρα μια ευκαιρία και υποστηρίζω αυτά που είπε ότι χρειαζόμαστε δηλαδή κάτι για την Ευρώπη. Αλλά επειδή κάποιες χώρες δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Θα πρέπει να πούμε πάσα ειλικρινία ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα ασαφές πεδίο. Θα πρέπει να είναι στόχος να αναπτύξουμε τα πιο υψηλά πρότυπα για την απόρριψη. Αυτό για μένα είναι, τι να σας πω, επιστημονική φαντασία. Θεωρώ ότι η στοχοθέτηση αυτή είναι σφαλμένη. Δεν υπάρχει σαφής ε, δήλωση για την ε, κατάργηση του άνθρακα και του πετρελαίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς οδηγίες για το προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε. Σαφείς αναφορές. Αυτές λοιπόν θεωρώ. Μία ερώτηση για την ενεργειακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Στο σημείο 15 στο σχέδιο αναφέρεται την ενεργειακή συνεργασία με τρίτε χώρες. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε το θέμα αυτό λίγο παραπάνω. Η κυρία Κόμπουλα Ναντρέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καλνιέτε. Η παρουσίαση σας ήταν ξεκάθαρη και είναι καλό που συνεχίζουμε τις συζητήσεις από αυτόν. Να σα ευχαριστήσω επίση για την ε, ο, παρουσίαση του κυρίου Σεύκοβιτς εδώ σήμερα, χτες, συγγνώμη. Όταν ε, προσθέτουμε το θέμα της ε, ανανεώσιμες, χρειάζεται μια ευελιξία στο δίκτυο παροχής ενέργειας, όχι μόνο αγωγή διασύνδεσης, περιφερειακή συνεργασία, αλλά και ευελιξία του δικτύου σε περιφερειακό και πιο ευρύ επίπεδο. Αναφερθήκατε όμως και στη βιώσιμη βιομάζα. Εξέτασα τα πρόσφατα έγγραφα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς εκπληρώνουν τους στόχους του οι διάφορες χώρες. Μόνο τρεις χώρες, η Σουηδία, η Εστονία και η Βουλγαρία, πληρούν τους, χώρες τους, τους στόχους τους αυτούς. Στη Φιλανδία είμαστε στο 35% ενώ ο στόχος είναι 38%. Μόνο η Σουηδία και η Λετωνία έχουν παραπάνω. Έξι χώρες ανέφερα, πέντε εξ αυτών εξαρτώνται πάρα πολύ από την βιοενέργεια. Και πολύ φοβάμαι ότι κοιτώντα την βιοενέργεια Κάποιοι ασκούν κριτική στην βιοενέργεια. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στο μέλλον να υπάρχει βιώσιμη αξιοποίηση της βιοενέργειας, να, υπάρχει μεν, αλλά να αξιοποιείται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβανόφσκι λέει ο πρόεδρος. Επίτροπε. Α, σε σχέση με την Επιτροπή Μπαρόσο 2, η βασική ανησυχία τότε ήταν πώς θα βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της φιλόδοξης κλιματικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ταχαίως μεταβαλλόμενης ατζέντα για την ενέργεια. Εκτίθενταν θέματα τιμολόγησης αλλά και περιβάλλοντος. Και με την κυρία και με την Κόνι Χέντιγκαρτ. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, ανάγκη εξέβρεσης νέης ισορροπίας. Το θέμα ήταν όμως να μην κοιτάξουμε το ETS, το σύστημα εμπορία εμπορίας λοιπόν, πριν από το 2020. Σε ό,τι αφορά τη θέση σε εφαρμογή το 2018-2019 θα πρέπει να είναι σαφής ότι δυσχεράνουμε τη θέση μας, ότι βελτιώνουμε. Δεδομένη στις ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς κρίνεται το στόχο της επανομιομηχανοποίησης στο 20% και όχι 16% και διακόπτει ο Πρόεδρος. Next speaker will be, oh, uh, Mr. Benstein. Κύριε Μπένστεν, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομε ερωτήσει για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η προτεραιότητα αυτή θα γίνει πραγματικότητα με νομοθεσία και στα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν είναι ένα συνεργειακό πόρο, αυτό το αναγνωρίζετε. Και συμφωνείτε. Όμω, πώ θα γίνει η χρηματοδότηση κάποιων projects που θα έχουν σχέση με την αποτελεσματική χρήση τη ε, ενέργεια στα πλαίσια του πακέτου μέτρων για επενδύσει. Κύριο Γιάβορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε να μα μιλήσετε. Για Ενεργειακή Ένωση θέλω να ρωτήσω. Έχουμε τους πέντε πυλώνε της πρόταση Εύκοβιτς. Πολύ ωραία όλα αυτά και για την οικονομία χωρί ε, άνθρακα. Πάντως, μετά το Συμβούλιο της προηγούμενη εβδομάδας, παρακολουθώντας τη συζήτηση για την ενεργειακή στρατηγική, έχουμε την εντύπωση ότι έχει γίνει μια στροφή προς ε, την πυρηνική ενέργεια και όχι ενώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι θα γίνει όσον αφορά την συγχρηματοδότηση και τις επενδύσεις. Γιατί έχουμε δέκα κράτη τώρα, το οποίο έχουν παρεραπενθεί στο δικαστήριο γιατί δεν έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα. Δηλαδή, Δέσμε μέτρα τέλο πάντων για την ενέργεια. Κύριε Καπετανουρή είναι η επομένη. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομα. Μόνο μία ερωτησούλα στον κύριο Επίτροπο για την κατανάλωση. Αυτό κατανάλωση, γιατί όταν ολοκληρωθεί η περίοδος αυτή θα έχουμε μια σύσταση τον Ιούνιο για το θέμα αυτό από την Επιτροπή. Τι γίνεται. Είναι δυνατόν να έχουν εκεί πρόσβαση οι μεμονωμένοι, οι μικρότεροι καταναλωτές. Ευχαριστούμε, φίλε το λόγο. Συμπαθάτε με που ήμουν τόσο αυστηρός για το χρόνο αγόρευσης, αλλά πρέπει να φύγει. Σε 7 λεπτά ο κύριος Επιτρόπος. Τι να σας πω, πού να τα απαντήσετε τώρα όλα αυτά που ρωτήσανε κύριε Επίτροπε. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε. Πρώτο, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος, δεν είμαι υπουργό στην Ισπανική κυβέρνηση και δεν υπεραμείνομαι καμιάς εθνικής πολιτικής. Αλλά κάνουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική προ όφελο και των 22 κρατών μέλων. Ένα αυτό. Δεύτερο, Όντω, οι τιμέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλές και σε κάποιε χώρε πολύ υψηλέ. Και είναι σαφέ ότι είναι υψηλέ αυτέ τι τιμές. Και αν συγκρίνει κανεί τι τιμέ των ανταγωνιστών. Το σχιστοδοτικό αέριο ότι οι Αμερικανοί πόσο κερδίσανε και, και στο... Τι τιμή σε τιμή έχουν Οπότε ποτέ δεν θα έχει φτηνή ενέργεια σε τον υπόλοιπο κόσμο η Ευρώπη. Γιατί έχουμε όλο ένα και λιγότερο ρηκτά καύσιμα στις περισσότερες χώρες. Έχουμε εξάρτηση από τις εισαγωγές. Και είναι στριμωγμένοι καταναλωτές και για αυτό ο σκοπός της Ενεργειακής Ένωσης είναι το να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές στην ενέργεια. Ενία αγορά. Περισσότερους προμηθευτές. Εναλλακτικά από το φυσικό αέριο να έχουμε το υγροποιημένο αέριο. Τα εφή δίκτυα, περισσότερες επιλογές κλπ. Πρώτα πρώτα επομένω και η καλύτερη πολιτική για μας είναι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Για κάθε 1% αύξηση αποτελεσματικότητας μειώνονται οι εισαγωγές κατά 2,6%. Πάμε τότε για το στόχο του 40% λέει ο κύριος Τούρμες. Είδατε, είδατε τι είπα. Με είδατε. Άντε, 2,3. Είναι μια αρχή. Οπότε είναι σαφές ότι για να μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια θα πρέπει να αναλυθεί ο τιμολογιακός μηχανισμός. Το κόστος, η ε, έμεση φόρη, η λυπή φόρη Πρέπει να δηλαδή πώς διαμορφώνεται η τιμή. Αυτό να αναλύσουμε. Και είπαμε να μην έχουμε ε, κατευθυνόμενο μηχανισμό διαμόρφωση των τιμών. Γιατί έτσι δεν μπορεί ο ένας να πολύ ενέργεια στον άλλο. Γιατί κάθε χώρα έχει άλλο μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών. Όμως, εάν κανείς καταργήσει ε, αυτές τις φίξ τιμές, θα πρέπει κανείς κάτι να κάνει για την ενεργειακή φτώχεια. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει στην Επιτροπή. Γιατί είναι πραγματικά ένα πρόβλημα στην Ένωση. Όχι μόνο στην Ισπανία. Παντού. Η αποτελεσματική χρήση ενέργειας είναι το καλύτερο, γιατί αφορά τα κτίρια, λιγότερη κατανάλωση. Και γι' αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοια στρατηγική χρηματοδότηση για τα κτίρια φιλόδοξες στρατηγικές. Και πολλές φορές θα πρέπει να κάνουν κάτι και να αλλάξουν εσωτερική νομοθεσία. Γιατί να μπορέσει να μονοθεί ένα κτίριο, να έχει διπλά παράθυρα, θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι διοκτήτε. Πολλέ φορέ είναι 40-50 και ο καθένα θέλει τα δικά του. Οπότε πολλέ φορέ η Διεθνή Νομοθεσία ζητεί ομοφωνία, οπότε δεν γίνεται έτσι. Επομένω θα πρέπει όλοι μαζί και στι 28 χώρε να προβληματιστούν, να σκεφτούν πώ θα υλοποιήσουμε Γιατί 80% είναι μία αποτελεσματική ακτήρια Και 40% της κατανάλωσης είναι από τα κτίρια. επομένω να δούμε πώς θα έχουμε αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα κτίρια του καλοκαίρι και το χειμώνα. Συνδυασμός μέτρων. Κυρίως κοινωνικής πολιτικής. Με συνεργασία περιφερειακών, αργών τοπικών κλπ. Αλλά ακόμα και έτσι θα συνοηθούμε και με την κυρία Τάισεν. Να μην έχουμε φίξ τιμές και από την άλλη μεριά να καταπολεμήσουμε την ε, ενεργειακή φτώχεια. Όλοι οι αρμόδιοι επίτροποι σε συντονισμό, συνεργασία και με εθνικές αρχές, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κανόνες καταναλωτών, όλους με όλους, με όλους, για να δούμε πώς μπορούμε κάτι να κάνουμε. ακόμα και για τον ευάλωτο καταναλωτή και την, ε, και την ενεργειακή φτώχεια, ούτε εκεί δεν έχουμε κοινό ορισμό. Ε, και αυτό θα πρέπει να ε, μας απασχολεί. Επίσης, κάποιος ρώτησε ναι, τι θα γίνει με το ίσο και τις αρμοδιότητες τις σχετικές για τους ρυθμιστές. Οπότε υπάρχουν πολλά ζητήματα εκεί και θα πρέπει να το επεξεργαστούμε το θέμα και θα προσπαθήσουμε τα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την καινούργια εσωτερική αγορά να δούμε πώς θα έχουμε ένα καινούργιο κανονιστικό πλαίσιο και να ενισχύσουμε το Acer να είναι ανεξάρτητο και να έχει αρμοδιότητες κανονιστικές ώστε να υποπτεύει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τους σχετικούς κανόνες και επίσης, κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό, να χειρίζεται και διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει να προσαρμοστεί το ΆΙΣΕΡ για του. για τις νέες πρωτοβουλίες, για κάποιο είδους ε, συντονισμό όσον αφορά τα κτίρια. Άρα ξανοίγονται πάρα πολλές δυνατότητες και ε, εναλλακτικέ για το ICER, εάν περιχαρακώσουμε τις αρμοδιότητες και επίσης έχουμε την καινούργια εσωτερική αγορά όπου θα διανοηθεί πολύ σημαντικό ρόλο το ICER όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα υποκαταστήσει τους εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Θα το ενισχύσουμε όμως το γιατί υπάρχουν πολλά θέματα και διασυνοριακές πρωτοβουλίες όπου δεν μπορούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να κάνουν τίποτα. Να, η αξία του κοινωτικού δικού. Α, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ψηλά είναι ο που έχουμε όσον αφορά τη συνάντηση των Παρισίων. Για το 2050 είπαμε 60% μείωση των εκπομπών. Γιατί 60%? Γιατί μπορούμε έτσι να το βοηθούμε στην αλλαγή του κλίματος των δύο βαθμών που θα έχει ανέβει η θερμοκρασία. Όμω δεν αρκούν οι δεσμεύσει που έχουμε σήμερα για τη συνάντηση στο Παρισίο. Μόνο η Ελβετία κατέχει κάνει για τι δεσμεύσει μόνο η Ελβετία, αλλά καλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καμία άλλη χώρα. Ο, λέμε το μόνο που κάνουμε, λέμε και λέμε όλοι να έχουν φιλόδοξες προτάσεις. Και έτσι όμως ε, δεν έχουμε ίσες ισόρους ανταγωνισμού. Προσπάθησαν πάντως πάρα πολύ σκληρά με τη είπα και τους άλλους εμπλεκομένους, ούτως ώστε όλες οι αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες να έχουν κάποιες φιλόδοξες δεσμεύσεις. Πριν τη συνάντηση των Παρισιών, το COP21. Γιατί έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια δυναμική διαδικασία. Δυναμική διαδικασία των φιλοδοξιών. Πρόκειται για εξελικτική διαδικασία, μια διαδρομή αν δεν φτάνουμε για τους δύο βαθμούς όταν φτάνουμε στη, στη συνάντηση των Περσίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ε, ε δεσμεύσει, αλλά υπάρχει αυτή η πορεία που έχει ξεκινήσει για προβληματισμό, ανάλυση και τελικά να καταλήξουμε σε κάτι. Να, ποια είναι η πρόκληση του αιώνα. Τώρα, τι γίνεται με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου και γιατί να μην βάλουμε και τιμή για το διοξείδιο του άνθρακα. Άλλο αγορά άνθρακα, άλλο φόρος άνθρακα. Υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ και κατά. Θα πρέπει να συζητηθούν στους, στα κατάλληλα επίπεδα. Τώρα έχουμε και την πιο αποτελεσματική αγορά άνθρακα του κόσμου. Δεν είναι τέλεια. Και μας είπε για τη σταθερότητα της αγοράς ο κ. Λεβαντόφσκης. Ξέρετε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Αν πάντως υπάρξει υποστήριξη για την ε, έγκαιρη εφαρμογή, καλώς αλλιώς θα μείνουμε στην αρχική μας πρόταση και θα συμμετέχουμε επικοδομητικά στην ανέβρεση καλής συμβαστικής λύσης. Πάντως θέλουμε σωστά μηνύματα για τις τιμές άνθρακα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βρούμε συμφωνία. Επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Τι γίνεται με το ανάνθρακα, το πετρέλαιο, την πυρηνική ενέργεια, το σχιστολιστικό αέριο. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το σωστό ενεργειακό μείγμα. Αλλά θα πρέπει να τηρούνται υψηλότερε διαγραφέ ασφάλεια είτε διαλέξει κάποιο την πυρηνική ενέργεια, είτε το σχιστολιστικό αέριο. Θέλει περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Επίση, αν κανεί διαλέξει τον άνθρακα, ε, να περιορίσει τι ε, εκπομπές εξουδίου του άνθρακα και να ενισχύσει την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Είναι σαφή η εικόνα τι θα πρέπει να γίνει στην κάθε περίπτωση. Με πλήρη σεβασμό του δικαιώματο του κάθε κράτου, να αναπτύξει το δικό του μείγμα πολιτική. Επίση, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειαζόμαστε ένα ανώτατο ποσό και θα πρέπει να έχουμε και μία παραγωγή ενέργειας εναλλακτική και χρειαζόμαστε υποστήριξη των ΑΠΕ, χρειαζόμαστε διασύνδεση, αλλά διαφορετικές πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση να ενισχύσουμε και στο μέλλον. Τώρα, για την αυτοκατανάλωση. Όταν είχαμε υποβάλει την ε, ανακοίνωση για την ε, ελληνική αγορά, η αυτοκατανάλωση και αυτοπαραγωγή ήταν από τα βασικά θέματα. Υπάρχουν όμως διαφορετικές ε, μορφές αυτοκατανάλωσης. Συνήθως έχουμε τέτοια κατανάλωση όταν οι μεμονωμένοι καταναλωτές ανανεώσιμων πηγών ενέργεια συνδέονται με το δίκτυο. Πάντω θα έχουμε στενέ επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να υποβάλουμε τις πρωτοβουλίες. Θα έχουμε γενικές συζητήσεις, θα βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά και θα υποβάλουμε τις πρωτοβουλίες μας σε πλήρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεσμεύομαι να έρχομαι όσο συχνά με αντέχετε κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την παρουσίαση, για την ανταλλαγή απόψεων. Πραγματικά αναμένεται έντονη νομοθετική δραστηριοποίηση στα θέματα ενέργειας και κλίματος. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα, πολύ σημαντικό επίσης θέμα, αποτελεσματική χρήση των πόρων και μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Παναγίτσα μου, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Uh, uh, as usual. Συνάδελφοι, ο συνήθως uh, μας ενδιαφέρει να παραμείνετε στην αίθουσα μέχρι το τέλος της σα. Αν παρόλα αυτά θέλετε να αποχωρήσετε, να το κάνετε ήσυχα και γόργα. Madame Kumpula Natri as well. Please. Κυρία Κουμπούλα Νάτρη και για σας ισχύει το ίδιο. Περνάμε στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Συντάκτης γνωμοδότης ο κύριος Μπένετεκ Γιάβορ. Η νομοθετική πρόταση με θέμα την κυκλική οικονομία που ονομάζεται και West Waste Package έχει αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να κατατεθεί νέα βελτιωμένη πρόταση. Η Επιτροπή ΕΜΒΗ συνεχίζει την ενασχόληση με την κυκλική οικονομία με τη μορφή η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Η έκθεση μας είναι σημαντική όσο περιμένουμε τη βελτιωμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Μπενεντέκ Γιάβορ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα πεντάλεπτο το πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε πολύ καλά και εύστοχα, συνεχίζουμε ε, το έργο μας υπό έκτακτες συνθήκες. Γιατί όταν ανέλαβα τη γνωμοδότηση είχαμε ήδη ε, το πακέτο για τα απόβλητα στην ανακοίνωση για την κυκλική οικονομία. Ώσπου να εκφωνήσω όμως τη γνωμοδότησή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε το πακέτο της. Υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα ε, της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας. Καταρχήν εκφράζουμε τις προσδοκίες μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβάλει τη βελτιωμένη της πρόταση, όπως είχε υποσχεθεί ο Επίτροπος Τίμερμας και ο Επίτροπος Βέλε. Ελπίζουμε μέχρι την τέλη του χρόνου να υποβληθεί επιτέλου αυτή η βελτιωμένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επιπλέον στη δική μας έκθεση της πρωτοβουλίας ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει τη βελτιωμένη της πρόταση που όμως δεν θα επικεντρώνεται μόνο στο σκέλος των αποβλήτων στην κυκλική οικονομία αλλά θα αναφέρεται και στην παραγωγή. Και θα δίνει περισσότερη έμφαση και στις νομικές πτυχές ε, της παραγωγής, του σκέλους της παραγωγής στην κυκλική οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό και το υπόβεθρο της έκθεσης. Εγώ συζήτησα με τους και ηγητές και έχω συμπεριλάβει στο σχέδιο γνωμοδότησης περισσότερες προτάσεις των πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό και θεωρώ το σχέδιο γνωμοδότησης ε, αντικατοπτρίζει σχετικά πιστά τις προτάσεις και απόψεις των πολιτικών ομάδων. Και εδώ να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Και να πω ότι ήταν πολύ εύκολο το έργο εξαιτίας της συνένεσης που διαπιστώθηκε σε πολλά θέματα. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης, Αναφερόμαστε στην ενέργεια και στην αποδοτικότητα των πόρων που αποτελούν τη βάση οικονομίας, της βιομηχανικής ανανέωσης, προκειμένου να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, αλλά και να οδηγηθούμε σε αυτή την επαναβιομηχανοποίηση, γιατί η ανανέωση βιομηχανική δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε όσο πιο φορά ανάπτυξη γίνεται βέβαια. Επίσης λέμε ότι μία φιλόδοξη νομοθετική πρόταση προσδοκούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε μία, ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους και ολοκληρωμένα μέσα. Δεν θέλουμε δηλαδή κατακαιρματισμένες προτάσεις, αψηφιδωτά θα σε ενό ψηφιδωτού, αλλά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Επίση, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πακέτο με πολιτική, αηφόρο πολιτική διαχείριση των υλικών, που συζητήθηκε ήδη από τη Βελγική Προεδρία του 2010, να επανέλθουμε σε μια πολιτική για την αηφόρο διαχείριση των υλικών. Τώρα, το θέμα των αποβλήτων είναι πολύ σημαντικό. και υπήρχε και στο αρχικό πακέτο για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία. Το ξαναθέλουμε. Επίσης ε, αναφέρουμε την, όχι μόνο τη διαχείριση αλλά την ε, χρήση, τη συντήρηση και την επαναχρησιμοποίηση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Επίσης να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και η προστασία του καταναλωτή. Βιομηχανικές ε, συνέργειες αναφέρονται επίσης στο σχέδιο της γνωμοδότησης χρήση υποπροϊόντων ε, ως πρώτη ύλη ε, στον οικονομικό κύκλο και επίσης υπογραμμίζουμε το ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης για να δοθούν ε, κίνητρα για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια κυκλική οικονομία. Και τέλος, χρηματοδότηση των προτάσεων. Και στην ανακοίνωση για την κυκλική οικονομία και στο νομοθετικό πακέτο που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε σωστή πρόταση για τη χρηματοδότηση. Αλλιώς δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τα μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος εισηγητής, ε, τρία λεπτά. Ο κύριος ε, Γκάμπους από το ΕΛΚ, είναι ο πρώτος ομιλητής. Θα είμαι σύντομο. Μεγαλύτερο Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο του και συμφωνώ μαζί του. Όντω μπορούμε να κάνουμε σε κάτι καλό όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ κακό το ότι αποσύρθηκε η δέσμη μέτρων. Αλλά, αλλά, θα πρέπει να βλέπουμε πραγματικότητα λίγο πιο αισιόδοξα ε, λέμε ότι με αυτή την έκθεση μπορούμε να συμπληρώσουμε την, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε ένα παγίδο στο τέλος της χρονιάς και έτσι μπορούμε να έχουμε πιο ψηλά τον πύχη για κάτι πιο πλήρες από την προηγούμενη ρύθμιση. Οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να περάσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων που είναι φιλόδοξη και πλήρες. Γιατί έχουμε τώρα την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή οικονομία που σημαίνει αυτό περισσότερες θέσεις απασχόλησης, περισσότερη στήριξη στις ΜΜΕ και συνειδητοποίηση του ότι χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα της κυκλικής οικονομίας που πάει παραπέρα από μια οδηγία που είναι απλώς για τα απόβλητα όπως είπε και ο εισηγητής. Να συνδέσουμε την παραγωγή δηλαδή με τα απόβλητα. Είναι ένα στίχημα αυτό, μακροπρόθεσμο, όσον αφορά την κατάρτιση για οτιδήποτε που αφορά τα επαγγέλματα στην κυκλική οικονομία. Καλά, έχετε και βελτιωσούλε στο κείμενο, όλα αυτά θα γίνουν με τροπολογίε. Είμαστε στη διάθεση του ΣΥΚΤ. Ευχαριστούμε. Σοσιαλιστές Δημοκράτες τώρα. Κύριε Κίρτον. Κύριε Κίρτον Τάνλη μάλλον, συγγνώμη. Έχει κάποια υποχρέωση και έφυγε η Περβόνς Μπερέσα και εμείς χαίρομαι πάρα πολύ θετικό το σχέδιο κειμένο. Ευχαριστούμε. Τον εισηγητή ήταν πολύ καλή η συνεργασία του μαζί μας. Ανοίξαμε όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Δούλευα για τον κύριο Ποτόνι, ξέρετε, πριν έρθω στο κοινοβούλιο ως ευρωβουλευτής. Οπότε ξέρω την υπόθεση αυτή. Και θεωρούμε ως πολιτική ομάδα ότι αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτως ώστε να έχουμε ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κοινωνική πολιτική και μιλάμε για δύο εκατομμύρια θέσει εργασία μπορεί να έχουμε τώρα. Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή και για το περιβάλλον και δυστυχώ, δυστυχώ υπήρξε απόσυρση τη πρώτα εκείνη. Όμω ίσω ε, δεν είναι και τόσο κακό γιατί εκείνοι που είχαν δεσμευθεί συνέχισαν τον αγώνα τους τόσο ώστε να φροντίσουν να μην είναι ζωντανή αυτή η ιδέα. Η βιομηχανία, τα κράτη-μέλη, από παντού, από όλη την κοινωνία των πολιτών ε, μας το είπαν αυτό το θετικό μήνυμα. Επίσης, θέλω μια φιλόδοξη στρατηγική, όχι μόνο για τα απόβλητα Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι για τα απόβλητα. Υπάρχει το οικολογικό σήμα, για κάποια απειρχαιωμένα προϊόντα, ρύθμιση, βιομηχανική συμβίωση και συνέργειες. Να προσεχθεί και αυτό μεταξύ των επιμέρους κλάδων και τομέων. Δούμε θα γίνει και με τις δευτερογενείς ή δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Το θέμα είναι τελικά η βιομηχανία να δημιουργήσει θέσει απασχόληση, αλλά και σε άλλου ε, τομεί, όπω η επεξεργασία των αποβλήτων. Βέβαια είναι και το θέμα η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης θα δημιουργηθούν, υγεία, υγιεινή και ασφάλεια ε, προβληματίζουν τους σχετικούς κύκλους αυτά. Κατάρτιση, υγεία λοιπόν και ε, ασφάλεια. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε με κάποιες τροπολογίες και ελπίζουμε ότι η αγαστή συνεργασία θα συνεχιστεί και με τις τροπολογίες. ήταν Σέρπα. Α, από ό,τι βλέπουμε συνεχίζεται τώρα και σκαρφουλώνεται ψηλά βουνά. δύσκολο. Φέντερλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και του ε, συναδέλφου, του ε, σκιώδε για την καλή συνεργασία. Και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Κατά βάση τα ίδια έχω να πω με αυτά που είπα και στη συνεδρίαση των ε, σκιωδών σε πιο κλειστό κύκλο. Πιστεύουμε ότι η γνωμοτότητα σε αυτή τη φάση είναι αρκετά στεναρή σε ό,τι αφορά την αντίδραση για τα απόβλητα και τις συσκευασίε. Τώρα έχουμε την, ε, απόσταση του πακέτου για τα απόβλητα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε στα θα γίνει και παραπέρα. Να μην να κοιτάξουμε μόνο τα απόβλητα, αλλά τι πόρου έχουμε στην κοινωνία που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιούνται με καλύτερο τρόπο για να υπάρχει καλύτερη αποδοτικότητα των πόρων. Επίση, θέσαμε διάφορα ζητήματα τα οποία είναι προβληματικά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία, ισορροπία μεταξύ αρμοδιοτήτων των εθνικών κρατών μελών και των όσων θέλουμε να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει κάποια σύγκρουση. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να μιλήσουμε και να ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε ότι κάποιες πολιτικές ε, θα πρέπει να προωθηθούν σε, ευρωπαϊκ... σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η ιδέα της εκτενούς ευθύνης του παραγωγού έχει δώσει μια τελείως καινούργια ανατροπία στη Σουηδία σε ό,τι αφορά τις συσκευασίε. Πριν από 15 χρόνια, στα μικρομάγαζα, υπήρχε πρόβλημα με όλα τα απόβλητα. Κάποιος έπρεπε να, να τα ε, μαζέψει, να τα κάψει επιπληρωμή. Και τώρα άλλαξε η νοοτροπία και πλέον ε, χρησιμοποιούνται ως πόροι τα απόβλητα αυτά. Και σε ό,τι αφορά την πρόθεση της οικονομίας και των θέσεων απασχόλησης. Σε κάποιες ε, περιπτώσεις η ανακύκλωση φτάνει μέχρι το 90%. Πρόκειται για ένα ισχυρό κλάδο και ε, ένα κλάδο για πολλές θέσεις απασχόλησης. Και αυτό προωθεί και κάποιες βασικές αξίες στην κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει και αντομικό τμήμα, βιομηχανικό τμήμα και αυτά να ενισχυθούν για να ενισχύσουν με τη σειρά τους και την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα καταθέσουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίες, αλλά θεωρώ ότι μια μεγάλη πλειοψηφία της ομάδας είχε πραγματικά προοδευτικές ιδέες. Και πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό το σημείο εκκίνησης για να ξανατεθεί το θέμα και να μπει να μπουν τα σημεία της ημερήσιας διάταξης της ατζέντα. Λοιπόν, πιστεύω ότι πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, επόμενους ομιλητές από την ΚΟΕ. Ο Λαφ Λάμσορφ που είναι και αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό το θέμα, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλες τις βασικές οικονομίες του κόσμου. Όταν μιλούμε για την κατανάλωση της ενέργειας, ένα θέμα πολύ συζητημένο, ξέρουμε ότι η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και η κατανάλωση πρώτων υλών μακροπρόθεσμα μπλοκάρουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Η Κίνα μάλιστα εξέπληξε για τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες με, την, με τους χοργούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Πρόσφατα όμως το πρόβλημα των αποβλήτων και της ε, υψηλής κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας ε, μπλοκάρει την οικονομία της Κίνας. Και με το περιβάλλον υπάρχει πρόβλημα. Ένας Αμερικανός οικονομολόγος ε, με πολύ περίεργο όνομα ε, δημοσίευσε ένα βιβλίο για την Κίνα και είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και σε σύγκριση με την Ινδία που έχει διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης η ενεργειακή κατανάλωση στην Κίνα είναι τριπλάσια από ό,τι στην Ινδία. Και σε σύγκριση με την Ευρώπη είναι εξαπλάσια η ενεργειακή κατανάλωση στην Κίνα. Οπότε τώρα το περιβάλλον και η ατμοσφαιρική ρήπαση, η μόλυση του νερού και η ρήπαση του εδάφους βάζουν τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και δημιουργούν και κίνδυνο για την κοινωνία. Μάλιστα στις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία των Κινέζων συμφωνεί ότι ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι όλο και πιο σημαντικός. Και γι' αυτό ο κόσμος δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον. Ακόμη και με κόστος την επιβράδυση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. Το περιβάλλον λοιπόν είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι σημαντικός και για την απασχόληση. Γιατί ο κλάδος της προστασίας ε, και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει ένα λόγο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ούτως ή άλλως ε, έχουμε ε, πάρει το κατήφορο στη μεταποίηση και μάλιστα πέρυσι δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο για τα 30 θριαβευτικά χρόνια του καπιταλισμού και πρόβλεψε τη, την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Αυτά στη δεκαετία του 60. Τώρα ακόμη και οι υπηρεσίε έχουν φτάσει στα όρια του. Οπότε να ζητούμε νέε ε, ευκαιρίε για θέσει απασχόληση. Και το περιβάλλον και η δημιουργία μια κυκλική οικονομία μπορούν να αποτελέσουν ε, τομεί ε, που θα δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία. Ευχαριστώ κύριε Σταμπουράνο. Συμφωνούμε 100% με τα όσα είπε ο κύριος ευχαριστούμε. Πάντως έχουμε και εμείς κάποιες ε, προτάσεις και θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο όσον αφορά τα, τα απόβλητα από εμπόριο και από βιομηχανία, οπότε εμείς θα κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες, τόσο ώστε να μην υπάρχει ανευθυνότητα και να υπάρχει ενεργειακή ανάκτηση από τα απόβλητα αξιοποίηση να έχουμε αυτό που λέμε καινοτομία γλωσσολογική στην Ιταλία και οπότε θα πρέπει να έχουμε έτσι κάποιες ε, πρώτες ε, ύλες και αυτές τις δευτερογενείς τις μη ε, ανανεώσιμες οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια μετακύληση του βάρους, του φορολογικού από την εργασία στα απόβλητα και στους πόρους και έτσι να έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής τα προϊόντα. Επίσης, θα προτείνουμε μία αλλαγή όσον αφορά τη διάρκεια της εγγύησης των ευρωπαϊκών προϊόντων. Και έτσι τα, τα διάφορα προϊόντα θα παλιώνουν ε, παλι, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλωσορίζουμε ασφαλώ τι προτάσει τη Ευρω... και η ιδέα για την μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων και το ότι υπογραμμίζονται οι πτυχέ τη ανταγωνιστικότητα χωρί να ξεχνάμε τι μικρομεσαίε. Σημειώνουμε τα διάφορα σχόλια που έγιναν εδώ σήμερα και στις προτάσεις σας κάνατε πολύ σωστά το σύνδεσμο, τη σύνδεση με το επενδυτικό πρόγραμμα που θα πρέπει να υποστηρίξει τα κρατημέλη προς τη μετάβασή τους για μια ε, κυκλική οικονομία. Όπως αναφέρατε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται επί μιας νέας πρότασης για την κυκλική οικονομία. Το νέο πακέτο θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης και μια αναθεωρημένη πρόταση για τα απόβλητα για να εγκριθούν όλα αυτά πριν τα τέλη του έτους για να συμπληρωθεί το έργο λοιπόν που έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι πολύ χρήσιμο να λάβουμε τώρα τα σχόλια από πλευρά του Κοινοβουλίου μέχρι το καλοκαίρι, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λάβει υπόψη της αυτά όταν οριστικοποιήσει, όταν τελειώσει τις προτάσεις της. Θα κοιτάξουμε όλες τις φάσεις του κύκλου. Η ιδέα είναι να συνδεθεί καλύτερα η διαχείριση των αποβλήτων με την επίτευξη κάποιων στόχων και προτείνουμε ενισχυμένη προσοχή στο σχεδιασμό των προϊόντων στη διευκόλυνση της ανάπτυξη αγορών για προϊόντα ανακύκλωση. Και το σχέδιο δράσης αναμένεται ότι θα είναι πάρα πολύ λειτουργικό, θα εστιάζεται ε, στα βασικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την κυκλική οικονομία σε όλες τις ε, αλυσίδες ε, αξιών και αυτό προτείνουμε να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα θητεία της Επιτροπής. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη και θετική επικοδομητική ορμή για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι το θέλουν και το θεωρούν μια ευκαιρία. Τέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο δράσης μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου και Ιουλίου. Σας ευχαριστώ. η ναι, κυρία Φαμπάρ εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Α, το περιβάλλον. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Μάλιστα, πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Μάλιστα. Ο εισηγητής λοιπόν τώρα, αν θα ήθελε να πάρει το λόγο να κάνει κάποια καταλητικά σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Βέβαια, τέλειο κείμενο δεν υπάρχει. Κάθε σχέδιο είναι βελτιώσιμο. Και επαναλαμβάνω, περιμένω με δημονία τις τροπολογίες των σκιωδών εισηγητών. Βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή σκέψης και πιστεύω ότι θα βρούμε κοινά σημεία. με ενημέρωσαν ότι αντί για τις 26 Μαρτίου που ήταν η αρχική προθεσμία για την κατάθεση προ... τροπολογιών, μπορούμε να προβλέψουμε νέα προθεσμία την 8η Απριλίου. Μια μικρή αναβολή για να προλάβουμε και να καταθέσουμε τροπολογίες και να το συζητήσουμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχουν έκθεση επίσης για τα υλικά για να συντανιστούμε οι δύο εισηγητές γνωμοδότησης ως προς τη διατύπωση και τις κατευθυντήριες γραμμές. Πάντως ε, ευελπιστώ ότι το οριστικό κείμενο θα είναι ικανοποιητικό για όλους και παραλαμβάνω ότι η κυκλική οικονομία είναι σε νευραλική σημασία ζήτημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους και να δημιουργήσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά μας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την εξάρτησή μας ε, από πρώτες ύλες. Ευελπιστούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το βελτιωμένο της ε, νομοθετικό πακέτο που θα πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ήσταν πολύ αποτελεσματικός γιατί με προλάβατε. Εγώ είχα σκοπό να πω ότι υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας μέχρι τις 8 Απριλίου, Άρα, τα είπατε εσείς. Πολύ ωραίο, είναι πολύ πιο σημαντικό να μας ενημερώνει απευθείας ο εισηγητής μας. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει τον Ιούνιο τους σε άλλους, οπότε χρόνος υπάρχει. Οπότε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών η 8η Απριλίου, όπως μας είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο 17, την εφαρμογή της οδηγίας, πολύ περίπλοκο το νούμερο, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ης Μαΐου του 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Για μας το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί Έχουμε κάποιες αρμοδιότητες για το copyright και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί και η έρευνα και η καινοτομία εμπίπτουν σε αρμοδιότητες της Επιτροπής Ήτρε και επίσης είμαστε αρμόδιοι και για την κοινωνία της πληροφορίας. Συντάκτης της γνωμοδότησής μας είναι ο Χωσέ Μπλάνκο Λόπες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω που με ορίσατε εισηγητή για αυτή την έκθεση. Πολύ σημαντικό το θέμα. Πολιτισμός, καλλιτεχνική δημιουργία είναι το τι είμαστε εμείς ακριβώς και αυτό που μας διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο κόσμο, μας στην Ευρώπη. Ο πλούτος και η πολυμορφία, η πολιτιστική είναι το πιο μεγάλο μας κεφάλαιο. Βέβαια μιλούμε και για βιομηχανία και οικονομική ε, δράση και μιλούμε για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Πάνω από 7 εκατομμύρια ε, να απασχόληση, πάνω από 2% ε, του ε, χώρου προϊόντος. Αυτά γίνονται, φανταστείτε, σε μια συγκυρία σοβαρή κρίση. Οπότε και αυτό το οποίο εμεί θα είναι να βρούμε ένα πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι αυτό που μας δίνει ταυτότητα ως κοινωνία και μας διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο κόσμο και γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο για οικονομική ε, ε, δραστηριότητα. Οπότε και αυτό το οποίο προσπάθησα σε αυτό μου το κείμενο είναι να προστατεύσω τη δημιουργία και την βιομηχανία στον τομέα τον πολιτιστικό. Γιατί έτσι θεωρώ ότι θα εξασφαλιστεί προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Πρόκειται για κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με τα ψηφιακά και επίση τα δικαιώματα των δημιουργών αφορούν τον πολιτισμό μα και από εκεί πηγάζει η δραστηριότητα η οικονομική, η ανταγωνιστικότητα αλλά και η απασχόληση γιατί εάν δεν έχουμε όμω κάποια αμοιβή δίκαιη δεν υπάρχει δημιουργία. Χωρί δημιουργία δεν υπάρχει και δικαιώμα, δεν έχει νόημα η προσβασιμότητα. Οπότε έχουμε πριν από 10 χρόνια τη σχετική οδηγία. Οπότε για τώρα πρέπει αυτή να αναθεωρηθεί οπότε επίση να διαπιστώσουμε ότι είχαμε από κάποιε μελέτε κάποιε πρόοδου. Και αυτό μα το λένε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και προκύπτει ότι η ψηφιακή αγορά ε, μπορεί να μας οδηγήσει σε σωστή αμοιβή των δημιουργών αλλά και σε αποτελεσματική και δίκαιη κατανομή των εσόδων στα πολιτιστικά και επίσης ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίε από την κατάτμιση τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση από αξιοποίηση από την οδηγία του 2014 να έχουμε αυτές τις εγκρίσει. Ε, ε, που αφορούν πολλούς χώρους, πολλά, πολλές χώρες και έτσι να μπορέσουμε να άρουμε τους ε, φραγμούς τόσο να υπάρχει πρόσβαση πέρα και πέρα από τα σύνορα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τίποτα όμως δεν γίνεται εάν δεν ε, μπορέσουμε να, να προστατεύσουμε αυτό τον κρίκο που αφορά τον ερμηνευτή, τον καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο πιο δυνατό κρίκος. Οπότε να έχουμε ένα πλαίσιο μετά τις διαπραγματεύσεις και να δούμε ότι χωρίς δημιουργούς δεν υπάρχει δημιουργία. Ούτε έχει νόημα η πρόσβαση σε έναν πολιτισμό, σε κάποια πολιτιστικά πλούσια και πολύμορφα. Τα ψηφιακά είναι προφανές ότι μας δίνουν καινούργια πρόσβαση και έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε νέες ε, επιχειρηματικές ε, πρωτοβουλίες. Όμως δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και τους κινδύνους. Πώς δηλαδή μπορεί κανείς να παρακάμψει τους κανόνες για τις δίκες αμοιβές. Και αυτό βλέπουμε κάθε μέρα. Άρα το πιο ευφιές, το πιο δίκαιο θα ήταν οποιαδήποτε αναθεώρηση για αυτό το θέμα να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας και επίσης να έχουμε ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο και έτσι να έχουμε ασφάλεια δικαίου αλλά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στον πολιτισμό. Και έτσι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας, τη δίκαιη αμοιβή στους δικαιούχου και επίση να υπάρχει βοήθεια από την ψηφιακή τεχνολογία που μπορούν να προσφεύγουν οι χρήστες και αυτό είναι ο στόχος του κειμένου που, που σας παρουσίασα. Ε, thank you much, ε, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιγητά. Ή σκιώδη Σιγητές τώρα. Η κυρία Βαλεάν, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω τον Ισίγητη για την γνωμοδότηση που μας παρουσίασε. Νομίζω ότι αποτελεί ένα εξαίρετο σημείο κίνηση για τι συζητήσει μας. Υποστηρίζω όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και φυσικά το στόχο, του στόχου που αναφέρει ο Θα καταθέσω παρόλα αυτά κάποιες ε, τροπολογίε για να εμπλουτίσω την γνωμοδότηση. και για να σχολιάσουμε κάποια από τα ζητήματα που ακούσαμε στη συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ιδιαίτερα κάποια ζητήματα γνωστά. τα οποία σίγουρα θα αναφέρει και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γνωμοδότηση. Ένα θέμα είναι το θέμα της εδαφικότητας, το οποίο αποτέλεσε ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να κάνει θεώρηση της ε, νομοθεσίας του δικαιώματος του δημιουργού. Και το θέμα της ε, φορητότητας είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ε, εξέβριση δεδομένων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά το επιστημονικό έργο, ένα παράλληλα να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα του, των ιδιωτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί σήμερα οποιοδήποτε που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι δημιουργός. Αλλά να φροντίσουμε ότι προστατεύονται και γνωρίζονται παρκώς οι αρχικοί δημιουργοί, οι αρχικοί συγγραφείς να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ο συνεχιζόμενος διάλογος και συνεργασία για το νομοθετικό πλαίσιο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών προκειμένου να μην υπάρχουν περιτά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά σε ό,τι αφορά θέματα copyright. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Νομική Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, ενημέρωση, ανανέωση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να περιοριστεί όμως το θέμα των ε, δικαιωμάτων του δημιουργού που αποτελούν τη βάση για την ε, δημιουργικότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, έχετε απόλυτο δίκιο που μας υπενθυμίζετε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η αρμόδια άλλωστε επιτροπή και ζήτησε έγκριση για την ε, υιοθέτηση της οδηγίας, μάλλον για την ενημέρωση της οδηγίας του 2001 σε ό,τι αφορά την ενημέρωση στις σύγχρονες πραγματικότητες. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστώ. από την Άλντε, ο κ. Κυριώτα Ταβιντάλ. Η προηγούμενη μήτρια από το ΕΛΚ ήταν. Τώρα η Άλντε έχει το λόγο. Ο κύριος Γκυράου Ταβιδάλ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την ισορροπημένη του γνωμοδότηση. Μπράβο. Η ο τομέας της ε, δημιουργίας και του πολιτισμού είναι σημαντικός και για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την κοινωνική ένταξη και την πολιτική πολιτιστική πολυμορφία. Και αυτοί οι κλάδοι εξακολουθούν να δημιουργούν θέσει απασχόληση παρά την κρίση. Βέβαια υπάρχει κατακαιρματισμό τη αγορά, δεν υπάρχει εναρμόνιση και έχουμε περιορισμούς, ε, Κάτι που αποδίζει την διασυνοριακή μερικές φορές πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία. Επίσης έχουμε κάποιες καταχρήσεις ε, στο διαδίκτυο μετά την οδηγία για το copyright του 2001. Το copyright είναι η ρεχοκοκαλιά της ε, πολιτιστικής πολιτικής, ε, στηρίζει τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την πρόσβαση στα έργα δημιουργού. Βέβαια πρέπει να προσαρμόσουμε την ανάγκες μας στις νέες συνθήκες της ψηφιακής αγοράς και να εξασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών φυσικά με, σε, με ικανοποίηση των προσδοκιών και των καταναλωτών. Χαίρομαι για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξυγχρονίσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το copyright, προκειμένου να προσαρμοστεί αυτό το πλαίσιο στην ψηφιακή εποχή. Η πολυδαφική αδιαδότηση είναι ένα σημαντικό βήμα για να ε, ξεπεράσουμε το κατακαιρματισμό της αγοράς, αλλά χρειαζόμαστε ισορροπημένες και ε, αποτελεσματικές λύσεις για να ξεφύγουμε τις ε, στενοπούς. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, νομικές ασάφειες. Κάποιες εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνουν ε, υποχρεωτικές. Και φυσικά οι εξαιρέσεις να μην αντιβαίνουν στην κανονική αξιοποίηση του έργου ή να μην θίγουν τα εύλογα και νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων. Σημαντικό αυτό το θέμα και για την έρευνα θα πρέπει να ληφθεί απόψη ε, στην οδηγία. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε το κατακαιρματισμένο σύστημα των εθνικών ε, συνεισφορών και να ε, βρούμε έναν τρόπο να μην τους δημιουργούς, όχι όμως εις βάρος των καταναλωτών. Επίσης, ξέρουμε, θέλουμε καλύτερη διαλειτουργικότητα του software και των τερματικών και να αποφύγουμε την δεσπόζουσα θέση στην αγορά που είναι εκ των ονοκάνευ προϋπόθεση για θεμητό ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια γιατί τηρήσατε το χρόνο σας. Ε, λυπούμε που πριν όταν είχαμε τον Επίτροπο σας διέκοψα, αλλά βιαζόταν ο Επίτροπος και δεν μπορούσα να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ τώρα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Θα ήθελα επί της αρχής να διευκρινίσω ότι και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση των δυνατικών δικαιωμάτων, αλλά να αναφέρω και μια άλλη πτυχή που δεν έχουμε ακούσει. Η κουλτούρα, η νοοτροπία της κοινή χρήσης ε, του μοιράζεστε και ότι θα πρέπει και ο δημιουργός να μοιράζεται τα αγαθά Αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να λεφθεί υπόψη πιο πολύ αυτή η πτυχή. Και για να επανέλθω στην ε, έκθεση επί της οποίας γνωμοδοτούμε, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε την προσέγγιση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο δίκαιο για τα, τα δικαιώματα του δημιουργού, το οποίο θα πρέπει να αντικατιστά τα εθνικά συστήματα. Αυτό είναι απαραίτητο για την ε, σαφήνεια και την βεβαιότητα, την νομική βεβαιότητα. Στη γνωμοδότηση υπάρχουν πολλά καλά σημεία, αλλά και πολλές ασάφειες. Για παράδειγμα, στην ε, παράγραφο 3. Θέλουμε η οδηγία 2001 96 να αλλάξει, αλλά για να ωφελήσει τους δημιουργούς. Και αυτό θεωρώ ότι δεν έχει αποτυπωθεί επαρκώς στο σημείο 5. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να παραμείνει. Και συμφωνώ με αυτά που λέει η Ιουλία Ρέντα στην έκθεση της. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι δεσμευτικές ε, όλες οι, όλες οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί προκειμένου να βελτιωθεί η νομική βεβαιότητα. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πτυχή που θα πρέπει να, προταθεί, να προσταθεί. Και το σημείο 7 είναι πολύ καλό για την διάσταση των αναπήρων χρηστών. Πολύ μας αρέσει αυτό. Κάποια λοιπόν στοιχεία θα πρέπει να βελτιωθούν και θα καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για τα σχόλιά σα. Άλλο κανεί. Να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο, τον κύριο Μάρκο Τσορέλο από την Γενική Διεύθυνση Connect. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους βουλευτές για όσα είπαν και για τόσα έκαναν μέχρι τώρα. Σε αυτή τη φάση δεν θα μακρηγορήσουμε γιατί παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, τα όσα συζητάτε και τη συμβολή των συναρμόδιων επιτροπών. Προς το παρόν. Η Επιτροπή απλώς επιβεβαιώνει όπως λέει και το πρόγραμμα του 2015, ότι πρόκειται να κατεβάσουμε κάποια πρόταση κάποια στιγμή φέτος για το copyright. Ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ποιους τομείς ακριβώς θα καλύψουμε και ακριβώς ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Όπως προείπα, στην ε, νομική επιτροπή σήμερα, φέτος, δεν θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα οποία είναι φραγμή στην ανάπτυξη της ψηφικής αγοράς σε σχέση με το copyright. Δεν αποκλείεται όμως το να καλύψουμε και θέματα άλλα από τα οποία μας ε, απασχολούν. Ίσως όχι όμως αναγκαστικά και με την φετινή πρόταση. Παρ' όλα αυτά θα δούμε ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε και θα επανέλθουμε με την νομοθετική μας πρόταση κάποια στιγμή φέτος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λέω πρόεδρος. Μπορούμε τώρα να επιστρέψουμε τον εισηγητή μας και να του δώσουμε την ευκαιρία για τα τελευταία σχόλια για σήμερα. Ευχαριστώ. Πριν τη συζήτηση σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους και ηγητές και με συναδέλφους που μου κοινοποίησαν τη γνώμη τους. Είχαμε κοινού κοινούς προβληματισμούς για το πώς θα διαμορφώσουμε μια ενιαία αγορά που θα προστατεύει, θα διευκολύνει την πρόσβαση στο, στην κουλτούρα και θα ε, ανταβίβει δίκαια τους δημιουργούς. Μερικές φορές έχουμε ένα ε, περίπλοκο παιχνίδι ισορροπιών και μερικές φορές ε, έχω ανάμεικτες συναισθήματα. Το θετικό είναι η επιθυμία να αναπτύξουμε τον κλάδο της του πολιτισμού γύρω από την ψηφιακή αγορά για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό θέσεων απασχόληση και τις καινοτόμες ε, βιομηχανίες. Το αρνητικό σκέλος είναι ο ο πειρασμός ε, να δημιουργήσω μια αντιπαράθεση μεταξύ δημιουργών και χρηστών και να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι μερικοί πρέπει να βγουν κερδισμένοι και άλλοι χαμένοι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η αντιπαλότητα και η αντιπαράθεση γιατί αν δεν προστατεύσουμε τους δημιουργούς δεν θα έχουμε περιεχόμενο, οπότε όλοι θα βγούμε χαμένοι. Οπότε θέλουμε δίκαιη αμοιβή των δημιουργών. Αυτό θα πρέπει να έχουμε πρώτα κατά νου. Βέβαια έχουμε και περιορισμούς ε, και φορητότητα, διασυνοριακότητα, πρόσβαση, στο περιεχόμενο και το καθεξής. Περιμένω τις τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ευκαιρία για να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε. Θα καταθέσω και εγώ τροπολογίες για μια εξαίρεση για ερευνητικού και εκπαιδευτικού λόγους και για το δανεισμό έργων σε ψηφιακή μορφή. Αλλά δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε μια ε, ψευτοσυζήτηση, εσφαλμένη συζήτηση μεταξύ καλών και κακών δημιουργών και καταναλωτών. Μερικές φορές αργήσαμε πολύ να προσαρμοστούμε στο αίτημα των χρηστών, γιατί στην αγορά της μουσικής ε, είχαμε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Επίσης, ε, χρήσιμο και το σύστημα της αδειοδότησης. Πολύ προσοχή λοιπόν, ε, γιατί ο τομέας αυτός δημιούργησε θέσεις απασχόλησης ακόμη και εν μέσω δραματικής κρίσης μερικές προτάσεις όπως αυτή του ενιαίου τίτλου θα είχαν αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα γιατί θα αποκλείσουμε έτσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την αγορά, θα μειώσουμε τον ανταγωνισμό και θα περιορίσουμε το ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ε, λογικές εξέλιξεις στην αγορά, όπως η πρόσβαση ενός συνδρομητή σε μια υπηρεσία όταν πραγματοποιήσει τα μεταξίδια. Ε, τι γίνεται όταν η μουσική είναι ευχάριστη, αλλά όχι ο στίχος, για παράδειγμα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία του επόμενου μήνε ε, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, εξετάζοντα την ε, προαναγγελθήσα μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα μελετήσω διεξοδικά τι τροπολογίε ε, και θα αναζητήσω μαζί σας το, την δίκαιη και απαραίτητη ισορροπία. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ χειρό το μήνυμα και πολύ στιβαρό. Τώρα εξαρτάται από τους συναδέλφους και από την νομική επιτροπή θα συμφωνήσουν με το μήνυμά σας που όμως θα επαναλαμβάνω ήταν ηχηρό, σαφέστατο και θα αποτελέσει τροφή για συζήτηση. Θα πρέπει όλοι να το καλοσκεφτούμε. Ολοκληρώσαμε το σημείο 17, περνάμε στο 18, τα διάφορα που δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω. Προσεχή συνεδριάσεις, καταρχήν προθεσμία για τις τροπολογίες. 25 Μαρτίου, αύριο στις 12 το μεσημέρι. Στο 17, συνάδελφοι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι λίγη διορία για τις τροπολογίες. Επόμενη συνεδρίαση, 14 Απριλίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Μεγάλη συμμετοχή και ραντεβού σε ένα μήνα περίπου στην επόμενη μας δηλαδή συνεδρίαση. Αλλά θα τα πούμε και σε άλλες ευκαιρίες πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.